Uh, so, good, good morning, everybody. Um, uh, sorry to be starting a bit late this morning. We were waiting for our rapporteur, Mr. Hatzimarkakis, to arrive. Καλημέρα σας. Μπορούμε να περιμένουμε να έρθει ο κύριος Χατσιμαρκάκης, αλλά μια και έχουμε και μια ομάδα της ε, Κομισιόν πρέπει να παρουσιάσουμε με τις προτάσεις ε, για την ε, πρόσβαση στο, στο, στον ιστότοπο στον ιστοτόπων οργανισμό του δημοσίου τομέα. Ο κύριος Χατζημαρκάκης ας έρθει πιο μετά, αλλά εμείς δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο. Ξεκινήσει η παρουσίαση της μελέτης λοιπόν ε, των επιπτώσεων από την Επιτροπή. Είναι πολύ γερή η ομάδα, δεν ξέρω ποιος θα κάνει την παρουσίαση. Ποιος είναι ο επικεφαλής της ομάδας της Επιτροπής, πείτε μας. Και άλλωστε πρέπει να πω ότι χαιρόμαστε πολύ που έχουμε τόσους πολλούς από εσά εδώ σήμερα. Καλημέρα σας. Προέρχομαι από την DG Connect. Ο συνάδελφος διπλά ασχολείται επίσης με την πρόταση, όπως και ο Γιώργος Φαντερ Λόιτεν, κύριος Κόμαρεκ και η κυρία Καρολίν Λεφλέρ από τις διοργανικές σχέσεις και μια νέα συνάδελφος ειδική ε, εθνική εμπειρογνώμων από τη Σουηδία, κυρία Έλμσχάιμερ και σας από τη Γενική Γραμματεία. Επίσης. Με χαρά βλέπω τόσο γερή ομάδα από την Κομισιόν, λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος. Σας ε, δώσουμε το λόγο σε εσάς για την παρουσίαση και μετά ακούμε και τις παρατηρήσεις παρουσίας των ε, μελών μας, των βουλευτών μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να περάσουμε λίγο χρόνο ε, για ε, τις διαφάνειες. Θα τις περάσω εντάχει και μετά θα ήθελα κυρίως να ασχοληθούμε με τις ερωτοαπαντήσεις γιατί θεωρώ ότι αυτές είναι οι πιο σημαντικές. Στις 25 Απριλίου θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων και θα έχουμε μαζί μας έναν εμπειρογνώμονα ο, οποίος θα σας εξηγήσει λεπτομερώς το θέμα της προσβασιμότητας η προσβασιμότητα δεν, είναι, δεν αφορά μονάχα ε, τα άτομα με ειδικέ ε, ανάγκες ε, ή τους αναπήρους. αναφέρεται σε ολόκληρη την κοινωνία, σε μια κοινωνία γυράσκουσα μιλισμονείται. Στην πρόταση αυτή βασιστήκαμε στην εσωτερική αγορά γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει κατακαιρματισμός των εθνικών εξειδικεύσεων όσον αφορά την προσβασιμότητα. Έχουμε τις διεθνείς ε, κατευθυντήριες ε, ε, γραμμές, τις οποίες οι περισσότερες χώρες πλέον υιοθετούν με κάποιες κατά το μάλλον ή των μεγάλες διαφορές και διαφοροποίησης. Η πρόταση που κάνουμε και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ τώρα είναι ότι πολλά μέτρα ε, βασίσαμε ε, στην ε, πάυση των διακρίσεων. Έχουμε επίσης και κάποια soft measures, ήπια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει η προσβασιμότητα ε, από όλους για τα δημόσια έγγραφα, ε, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει ε, και που θέλουμε. Και άλλωστε η αγορά δεν προτείνει τις φθηνές και σωστές λύσεις έτσι ώστε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Ε, υπάρχουν ε, κάποιοι ιστότοποι ε, για τους οποίους υπάρχει καλή προσβασιμότητα και θέλουμε το spillover αποτέλεσμα να είναι σημαντικό. Η παροχή πρέπει και στους ε, προμηθευτές αλλά και στους, ε, στα νοικοκυριά να δίνουν ε, καλή υπηρεσία. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε δύο κατηγορίες κρατών μελών. Τα κράτη τα οποία ήδη έχουν νομοθετικά μέτρα και γενικότερα μέτρα τα οποία αφορούν το, το πρόβλημα αυτό. Είναι 21 χώρες μέλη, 21 χώρες μέλη Έχουμε όμως πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις Και πρέπει να πω ότι τα, οι νέοι ιστότοποι που θα οικοδομηθούν βάσει των νέων αρχών ε, δεν θα κοστίζουν πολύ, θα είναι πιο φτηνά από τα, οι προηγούμενοι ιστότοποι. Ε, μετά έχουμε τις χώρες οι οποίες δεν έχουν καμία ε, πρόσβαση ε, και πρέπει να πω ότι τα ωφελήματα από την ε, γενικευμένη επιγραμμικότητα ε, είναι πάρα πολύ μεγάλα, ειδικά για τις ε, υπηρεσίες που και τώρα, αλλά που στο μέλλον κυρίως θα είναι διαθέσιμες μονάχα επιγραμμικά, η κατάσταση είναι πολύ καλή. Θα υπάρξει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μικρός διασυνοριακός ανταγωνισμός λόγω ακριβώς των διακυμάνσεων και των διαφορών που υπάρχουν στις εθνικές αρχές. Δηλαδή μπορεί ε, μία χώρα ε, να ε, είναι ας πούμε πάροχος για, τις, για τα Υπουργεία της Ε, ενώ ταυτοχρόνως λέει ότι ο πάροχος θα πρέπει ε, να υποβάλλεται ε, σε εθνικές εξειδικεύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι κάπως μειώνει τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ. θέλετε κυρία συνάδελφε να ξεκινήσετε με τις ερωτήσεις ή θέλετε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση κύριε Χατζημακακάκη. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εισηγησή της. Είναι προφανές τι έχουμε εδώ, αλλά πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, συλλάβουμε το σύνολο του προβλήματος, γιατί πολλοί κόσμος έχει περιορισμένες δυνατότητες, όπως ας πούμε η τυφλή. Οπότε είναι δύσκολο κανείς να επισκεφθεί και έναν ιστότοπο δημόσιο οργανισμού που είναι πάρα πολύ σημαντική λειτουργία που επιτελούν για αυτά τα πρόσωπα. Κοιτάξτε, για να καταλάβετε τι εννοώ, να σας πω τι ισχύει ας πούμε για, για το δικό μου ιστότοπο, τη δική μου ιστοσελίδα. Ακριβώς εξεργαζόμαστε με τους συνεργάτες μου ε, την τη, τη, δική μου στο σελίδα για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε αυτούς που έχουν περισμένες δυνατότητες. Οπότε θα κάνουμε και κάποιο είδου ε, επίδειξη να καταλάβετε τι εννοούμε. Γιατί ακριβώς αν κανείς δεν είναι τυφλός δεν μπορεί να καταλάβει τα προβλήματα των τυφλών. Θα πρέπει μένως κατά κάποιο τρόπο να αποκατασταθεί η έλλειψη της όρασης σε αυτά τα πρόσωπα. Και έχουμε ένα σωρό τομείς όπου όλα αυτά έχουν σημασία. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το δίκαιο της ιστορικής αγοράς. Ε, και εδώ πέρα συντρέχουν και, και άλλες διατάξεις όπως ας πούμε ε, το, το θέμα του πώς το δίκαιο καλύπτει την ισότητα γιατί υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές ε, λειτουργίες, οπότε θα πρέπει η Επιτροπή μας να ασχοληθεί και προς αυτή την κατεύθυνση να προχωρήσουμε επί τη βάση της προτάσεως που έχουμε στα χέρια μας και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε το οποίο ε, να είναι και φιλόδοξο ε, και ολοκληρωμένο. Ο πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως. αυτό το οποίο είπαμε πρόκειται να το δημοσιεύσουμε, να το δημοσιοποιήσουμε, τόσο ώστε να διαδοθεί. Τώρα υπάρχει κάποιο άλλο και ο για του σοσιαλδημοκράτε. Τέλο πάντων, κάποιο θέλει το λόγο. Α, ο κύριο Τασκόφη είναι εδώ. Κύριε Τέλο είμαστε πολλοί οι οποίοι ενδιαφερόμαστε εδώ παρόντε και μπορούμε να λάβουμε το λόγο. Πρώτα-πρώτα ένα μεγάλο μπράβο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ αξιέπαινο αυτό ω ε, εγχείρημα και πρώτα-πρώτα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι δυνατότητε ε, που υπάρχουν για εξέλιξη, για ανάπτυξη, ε, να δούμε όλου αυτού που περιθωριοποιούνται, γιατί ακριβώ δεν είναι θέμα έλλειψη δυνατοτήτων, καμιά φορά είναι και θέμα ηλικία. Όταν μιλούμε για τα ψηφιακά, θα πρέπει να δούμε πώς θα βγουν όλοι κερδισμένοι. Γιατί εδώ και μια διετία ασχολούμαι με το ζήτημα και είχα και έναν ιστότοπο στην Πολωνία, ούτω ώστε να είναι συμβατό με τους πάντες και κάποιοι που είναι πάρα πολύ ειδικοί μου άνοιξαν τα μάτια και κατάλαβα ότι πρέπει να βρω μια λύση ούτως ώστε να βγαίνουν όλοι κερδισμένοι και τελικά να υπάρχει μια ιστοσελίδα όπου στο διαδίκτυο να λειτουργεί αυτή στο σελίδα έτσι ούτως ώστε ε, ας πούμε εμείς μηχανές αναζήτησης ε, όλοι να μπορούν να, να δουλέψουν. Οπότε έτσι θέλουμε να, να προβληθούμε στο διαδίκτυο, θέλουν οι δημόσιοι οργανισμοί επίσης να προβάλλονται ε, οπότε και τους αυτούς μας ωφελούμε αλλά και τον άλλο κόσμο για αν το φροντίζουμε αυτό. Ανακύπτουν εδώ διάφορα ερωτήματα. Δεν, δεν θέλω να επικρίνω. Απλώς ε, έχω κάποιες απορίες. Πρώτα πρώτα, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Και εδώ ανακύπτουν κάποια ερωτήματα διότι νομίζω ότι ε, η οδηγία προετοιμάστηκε εδώ και κάποια χρονάκια. Επομένως θα πρέπει να ληφθούν τώρα υπόψη και κάποιες φρέσκες πρόσφατες εξελίξεις. Ας πούμε, υπηρεσίες για επιχειρηματίες, όπως ας πούμε η καταχώρηση μητρώου μιας εταιρείας. Ξέρω ότι υπάρχει κατάλογος, λίστα που προσαρτάται σε παράρτημα, αλλά θα πρέπει να καλύψουν και κάποιες υπηρεσίες οι οποίες δεν αναφέρονται εκεί. Πολλά είναι τα ερωτήματα, πολλά παραδείγματα μπορούσα να σας πω ας πούμε, καταχώρηση σε κάποιο μητρό πανεπιστημίων. Αυτό το γράφει. Δεν γράφει όμως για παιδικούς σταθμούς, ας πούμε. Ή γράφει για ε, κάποια δημοτικά σχολεία. Γιατί να περιζόμαστε ε, στο να αναφέρουμε μόνο τα πανεπιστήμια, γιατί μόνο για τα κρατικά πανεπιστήμια, ε, γιατί όχι και τα ιδιωτικά. Να, επομένως ένα σωρό ερωτήματα Βεβαίω θα πρέπει να επικαλεστούμε και την εθνική μας εμπειρία και έτσι να διευρύνουμε στη βάση το πεδίο εφαρμογή του ευελινικία της οδηγίας. Άλλο θέμα είναι το γιατί δεν υπάρχει μια πιο οριζόντια προσέγγιση. Δεν λέει τίποτα εδώ για τους δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών του δημοσίου, γιατί όταν λέμε για προσβασιμότητα, τότε ε, θα πρέπει να καλυφθούν και αυτές οι περιπτώσεις, ακριβώς όπως των δημοσίων διαγωνισμών προμηθειών. Και θα πρέπει τουλάχιστον να αναφέρουμε και αυτούς τους τομείς και αυτές τις δραστηριότητες για να έχει πιο οριζόντιο χαρακτήρα το κείμενο. Δεν είμαι ειδικό, αλλά με ενημέρωσαν κάποιοι ειδικοί και από ό,τι κατάλαβα θα πρέπει όσον αφορά τα πρότυπα να καταφέρουμε να υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό πρότυπο. Πάντως η οδηγία εδώ, το κείμενο παραπέμπει στα πρότυπα του ISO. Εκεί πρέπει όμως κανείς να πληρώσει. Ενώ υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί προτύπων όπου δεν χρειάζεται να καταβληθούν χρήματα. Ξέρω ότι αυτό είναι ειδικό θέμα, αλλά κάπως να το λάβουμε υπόψη. Είμαι ο συντονιστής του ΕΛΚ για την Συνταγματική Επιτροπή. Πάντοτε εξετάζω τις κατεξιοδότησες πράξεις, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει τελικά να είμαστε πιο ακριβείς και θα πρέπει κάθε φορά να εξασφαλίζουμε το ότι γίνεται ορθή χρήση αυτού του διαδικαστικού μέσου των κατεξιόδων πράξεων. Επομένως, να προσέξουμε τι γίνεται και με το παράρτημα και να φροντίσουμε να μην έχει απαρχιωμένο χαρακτήρα το κείμενο, το νομοθέτημα. Νομίζω ότι αυτό το νομοθέτημα για την προσβασιμότητα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε με τον τρόπο που είπα και μεγάλη μου χαρά να μου κάνει ένα φροντιστήριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί σας είπα δεν είμαι ειδικό ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που έχετε τόσο πολύ ασχοληθεί με το θέμα αυτό και το έχετε μελετήσει. Έχετε συμβάλλει πολύ. Κυρία Στάιλερ, για να δω, ο κύριος Γκάθο δεν είναι εδώ. Εκπροσωπείτε εσείς τους σοσιαλδημοκράτες, έτσι δεν είναι σήμερα. Η κυρία Γκέπχαρτ όμως είναι εδώ. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα που εσάς σας ενδιαφέρει πολύ. Μήπως γίνετε εσείς όδης τελικά. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους άλλους ομιλητές όταν έγινε ο λόγο για την ε, νηστότοπο, πρέπει να πω ότι και εμένα με έβαλε σε σκέψεις, γιατί καλό είναι να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές εμείς οι βουλευτέ, να μαθαίνουμε ένα από τον άλλον. Στο Ρωμένο Βασίλειο, όταν άρχισαμε να ασχολούμαστε με του τοπούς και άρχισα και εγώ να ξανασχεδιάζω το δικό μου, αρχίσαμε να βλέπουμε ε, δυνατότητες για επικοινωνία και νέο σχεδιασμό και νομίζω ότι είναι θετικό. Επίσης ε, μιλάμε για δημόσιες προμήθειες στην Επιτροπή μας πολύ συχνά και έτσι ήθελα να πω ότι είναι ενδιαφέρον το ότι τίθεται το ζήτημα αυτό, η προσέγγιση δηλαδή ως προς τον, τον τομέα των δημοσίων προμηθειών και την εφαρμογή του εδώ. Και όταν μιλούμε για ευέλτιστες πρακτικές εμείς ως ευρωβουλευτές, ουσιαστικά κοιτάμε και ποια είναι τα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται στην πρώτο καθεδρία. Γιατί μπορούμε πάλι από αυτά να διδαχτούμε, αλλά και να διαδώσουμε τη γλώσσα αυτή και τις πρακτικές. Λόγος έγινε βέβαια και για προδιαγραφές και θεωρώ ότι είναι και αυτό σημαντικό. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τι ε, γνώμη έχετε ως προς το θέμα, όχι της μόνο της προσβασιμότητας που συζητούμε, αλλά γενικά της πρόσβασης στα μέσα μεζικής ενημέρωσης ή τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πρόσβαση σε μια πληροφορία. Αν το δούμε λοιπόν σε μια ευκαιρία μέσα σε ένα κλίμα που αντιμετωπίζουμε αυτή την εποχή και την ε, δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες που προσφέρονται, χάρη στην ε, πρόταση. Γιατί ήταν ε, συνθλιπτική η πληροφορία ότι 40% λιγότερο του 40% των ευρωπαϊκών ιστοτόπων είναι προσβάσιμοι. Εμείς προσπαθούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχουμε πολύ ψηλότερα ποσοστά. Δεν ξέρω αν έχετε ε, ξέρω ότι είναι ίσω λίγο σκληρό έτσι όπω το ζητάω, αλλά μπορείτε ας πούμε, να μα πείτε ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κράτη τα οποία δεν κάνουν καλά τη δουλειά του σε αυτό το θέμα. Και έχουν ε, τι κακέ επιδόσει. Υπάρχει, α πούμε, κάποιο κακό μαθητή που πρέπει να καταγγείλουμε. Και επίση ε, θα επαναλάβω ότι χρειάζεται να μοιραζόμαστε τι βέλτιστε πρακτικέ εδώ στο Κοινοβούλιο. Ραφέλ, Ίσως με το website μπορείς να μας ε, δείχνεις και με την επόμενη συνεδρίαση πάλι και ο κύριος Χατζημαντρικάκης ασφαλώς που έχει ένα υποδειγματικό νομίζω ιστότοπο, θα μπορούσαν να μας δείξουν, να μας δώσουν ε, ε, το παράδειγμα. Κύριο Σέγκστρομ. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με όλους τους προγραλήσαντες. Πολύ καλό, πολύ σπουδαίο, ενδιαφέρον, ασφαλώς πρέπει κάτι να κάνουμε. Ιδιαίτερα Θέλω να συμφωνήσω με τον κύριο Ταρκόφσκι που αναφέρθηκε στις προδιαγραφές, γιατί είναι πολύ σημαντικές. Όσο πιο τυποποιημένη γίνεται η προσβασιμότητα, τόσο πιο εύκολο θα είναι, τόσο πιο καλό θα είναι, γιατί υπάρχουν και πολλά διαφορετικά συστήματα. Συστήματα τα οποία δεν λειτουργούν πάντα το ίδιο καλά. Ίσως λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε προς περισσότερη τυποποίηση. Γι' αυτό οι προδιαγραφέ είναι καλέ. Διαφορετικά αντιμετωπίζουμε μια. Θα, θα βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση, γελία κατάσταση. Γιατί αν, α πούμε, έχουμε μια οδηγία η οποία λέει ότι θα πρέπει ο καθένα να ακολουθεί προδιαγραφέ, ε, αλλά ταυτόχρονα θα επιβάλλει ένα τέλο για τη χρήση των προδιαγραφών, των υποχρεωτικών αυτών προδιαγραφών, θα είναι, πιστεύω, παραλογισμό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ταυτόχρονα όπως είπαμε, ο στόχος είναι η εναρμόνιση, η ευαλτίωση της ποιότητας, η νομοθεσία με τη μορφή της οδηγίας μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά στην προκείμενη περίπτωση έχουμε και τα τεχνολογικά, τα τεχνικά μέσα που μπορούν να βοηθήσουν στην επικοινωνία, στην εναρμόνιση καλύτερα της επικοινωνίας. Και έτσι αναπτύσσονται διάφορες λύσεις από τα κράτη-μέλη που πιστεύω θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, να δημοσιεύονται οι τεχνικές λύσεις αυτές με, τον, ε, ε, με, το, με τη μορφή του open source, να είναι προσβάσιμα δηλαδή στους πάντες, για να βελτιώνονται, για να διαδίδονται πολύ περισσότερο. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το open standards, τις δημόσια προσβάσιμες, τις προσβάσιμες από το κοινό προδιαγραφές. Αυτό νομίζω πρέπει να το ενθαρρύνουμε. Η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται σε όρους open source. ο πρόεδρος. Εγώ είμαι σκιώδη σου, οπότε να τα πω εγώ. Είναι ένα θέμα το οποίο και εγώ παρακολουθώ εδώ και αρκετό καιρό. Κύριο μέλημά μου εδώ είναι όχι ότι δεν πρέπει να το προωθήσουμε και με πολύ θετικό τρόπο, αλλά το πώς θα το καταφέρουμε. Χωρίς να θέλω να σας φέρω καμιά ψυχρολουσία. Ας δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη. και μήπως υπάρχουν και καλύτεροι τρόποι να τα καταφέρουμε. Γιατί στην αξιολόγηση ε, λέγεται ότι σχετικά ε, πρόωρα απορρίψατε την ιδέα του ενδοτικού δικαίου ε, και ότι μπορεί να υπάρξει, ότι διαπιστώνεται κατακαιρματισμό της αγοράς κτλ. Ναι, κατακαιρματισμό της αγοράς υπάρχει, επειδή έχουμε να κάνουμε με υπηρεσίες που είναι ιδιαίτερες υπηρεσίες κρατικές, δημόσιες των κρατών μελών, με τη δική τους ορολογία, με τις συνθήκες που διαφέρουν ριζικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Γιατί είναι και διαφορετικές, διαφορετική ρυθμή της εξέλιξης. Άρα θα πρέπει να διαρωτηθούμε πόσο αποτελεσματικό, προϊόν θα προσφέρει αυτό. Έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέσα να ξεκινήσει διαδικασίες επί για κάθε κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ε, προσφέρει ε, ευχερός προσβάσιμο ε, ιστότοπο για κάθε πανεπιστήμιο και κάθε δημοτική αρχή. Γιατί είμαι πεπισμένος ότι θα μπορούσα να πείσω με μία μικρή διατριβή που θα έλεγε ότι υπάρχουν προδιαγραφές, θα πρέπει να προωθηθούν κοινέ προδιαγραφές, η διαλειτουργικότητα, συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που υπόθηκαν εδώ. Επίσης, διατάξεις που ισχύουν και που αφορούν την παρακολούθηση, επιτήρηση και που πρέπει να τηρηθούν, γιατί και η εξωτερική πίεση η εξωτερική πίεση από τις οργανώσεις των χρηστών, των πολιτών στα κράτη-μέλη θα είναι ασφαλώς πολύ ισχυρός παράγων και μοχλός για την πρόοδο. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ιδέες και τους πόρους της θα μπορούσε να τους αφιερώσει στον προσδιορισμό οροσίμων για την ε, προσβασιμότητα. Περισσότερο παρά τη συλλογή των δεδομένων. Και έτσι τα κράτη-μέλη και κυρίως αυτά τα οποία ε, ε, κοιτάνε και τα δημοσιονομικά πιο πολύ, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να δουν το συμφέρον αυτής της ιστορίας με μια πλατφόρμα που θα μπορούσε να ξεκινήσει να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη μέσω ίσως δημόσιων προμηθειών. Βέβαια εδώ έχουμε νέα οδηγία, έχουμε νέα εργαλεία για τις δημόσιες προμήθειες, ώστε να ε, ε, ενθαρρύνονται οι δημόσιοι ε, φορείς ή λειτουργοί στην αναζήτηση πιο εφάνταστων και δημιουργικών μέσων για τις δημόσιες προμήθειες, για τις προκηρύξεις, άρα μπορούν να αξιοποιήσουν και αυτό το μέσον. Και επίσης, αν κοιτάξουμε τον ορίζοντα 2020 και τη χρηματοδότηση μπορεί να προσφέρονται σε τέτοιου είδου ε, είναι ε, πιθανό να βρούμε λύσεις καλές, γρήγορε, αποτελεσματικέ πολύ περισσότερο από ότι εάν αυτή η νομοθετική πρόταση, η οποία ασφαλώς θα χρειαστεί χρόνο πολύ και διαπραγματεύσει στα κράτη-μέλη, ε, θα χρειαστεί για να... ή θα, θα φέρει, τι αποτέλεσμα θα φέρει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει και βεβαίως να μας δοθεί ευκαιρία να αξιολογήσουμε την ε, μελέτη επιπτώσεων, αλλά δεν ε, βλέπω πουθενά την διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων. Και όπως είπα, δεν έχω καμιά αντίληση προς το να επιτευχθεί πραγματική ουσιαστική πρόοδο στην υπόθεση αυτή. Έχω εργαστεί και για τα θέματα της οικουμενικής υπηρεσίας προσωπικός, υπάρχει, για τις τηλεπικοινωνίες υπάρχει νομική βάση, μπορούμε να επιβάλλουμε τη διαλειτουργικότητα στις, ε, στους ε, παρόχους των τηλεπικοινωνιών. Δεν είμαι κατά, δηλαδή απλώ δεν είμαι πεπισμένο ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Βέβαια, εσεί μπορείτε να έχετε άλλα επιχειρήματα και να με πείσετε για το αντίθετο αλλά ίσως καλό θα ήταν να εξεταστούν οι εναλλακτικέ και ίσως θα μπορούσε ο εισηγητής να μας βοηθήσει σε αυτό. Θέλει κανείς άλλο το λόγο, παρακαλώ. Κυρία Φερχαΐεν, ε, πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και σωστό να επιδιώκουμε κάθε διευκόλυνση και ελευθερία ως προς την πρόσβαση, την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο. Απλώς δεν είμαι βεβαία ότι μπορεί να το επιτύχει με αυτή την νομοθετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολλά τα ασαφή σημεία, είναι πολλές οι προτάσεις για τα κατεξουσιοδότηση πράξης που προβλέπονται στο έγγραφο. Η δε συγκεκριμένη ε, εφαρμογή, η ο τρόπος εφαρμογής υλοποίησης, οι υποχρεώσεις που θα επιβαρύνουν τα κράτη-μέλη, αλλά και ε, μέσα στα κράτη-μέλη τις τοπικές περιφερειακές αρχές, δημοτικές αρχές κτλ. Είναι κάπως ασαφής έως ανύπαρκτες. Γι' αυτό λοιπόν και επειδή με ενδιαφέρουν και οι προδιαγραφές και υποστηρίζω τις ιδέες σας σε, πολλές, σε πολλά σημεία, ότι χρειάζεται αυτή η τυποποίηση, οι προδιαγραφές, αλλά πάνω απ' όλα η διαλειτουργικότητα, ώστε διαφορετικές τεχνολογικές προσεγγίσεις να είναι δυνατόν να, να συνδυάζονται, προκειμένου να λειτουργήσει ένας ιστότοπος. Θα έλεγα για τον τομέα των προμηθειών, παραδείγματι, όπου έχουμε να κάνουμε κυρίως με τον επαγγελματικό τόπο, ε, τομέα. Είναι πολλές ε, οι δυνατότητες και για επαγγελματική αποκατάσταση κάποιου ε, που ενδεχομένως έχει μια αναπηρία ε, και μπορεί να απασχοληθεί ε, χάρη σε ειδικέ τεχνολογικές δυνατότητες. Και εδώ έρχεται το ζήτημα της διαλειτουργικότητας, ότι δηλαδή δεν πρέπει η κάθε ιστοσελίδα να είναι προσβάσιμη με τον ίδιο τρόπο, αλλά πρέπει να είναι προσβάσιμη με την χρήση της ε, ίδιας ειδική τεχνολογίας που θα χρειαζόταν ενδεχομένω. Ευχαριστώ. Κυρία Ρούλε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι εάν ε, άλλα ε, ε, άλλοι τομεί, άλλε υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν άλλου φακέλου όπω τι ηλεκτρονικέ δημόσιε προμήθειε αναμείχνονται στην υπόθεση αυτή. Γιατί είναι πολύ δύσκολο για μα να πείσουμε τα κράτη-μέλη μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει προσδιοριστεί να υλοποιήσουν ε, τι υποχρεώσει αυτέ. Και δεν βλέπω κανένα νόημα να προσθέτουμε εκ των υστέρων κιόλα κάτι το οποίο δυσκολεύει ακόμη περισσότερο μια προσπάθεια που ήδη είναι αρκετά επώδυνη και δύσκολο να υλοποιηθεί. Επομένω, ε, και επειδή ξέρουμε ότι πολλές φορές ε, χρησιμοποιείται ως ε, λιδία λίθος θα έλεγα το ζήτημα των δημοσίων προμηθειών από ορισμένε υπηρεσίες επιτροπής, καλό θα ήταν να το αφήσουμε χωριστά, να μην το αναμέξουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χατζημαρκάκη, να απαντήσει η Επιτροπή πρώτα και μετά να σας δώσω εσάς το λόγο για να κλείσετε. Είναι και ο κύριος Μάντερς εδώ για το επόμενο θέμα. Μας πιέζει λίγο ο χρόνος, αλλά είναι σημαντικό, θα τα ακούσουμε. Η Επιτροπή λοιπόν πρώτα, για να απαντήσει παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω στο ε, θέμα του πεδίου εφαρμογής, το οποίο ε, είναι σημαντικό. ε, καταλήξαμε στη διαφάνεια που είδατε και στα 12 σημεία τα οποία στην ουσία είναι το αποτέλεσμα ε, το, του ηλεκτρονικού benchmarking ε, που κάναμε για το τι μπορεί να είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμο. Είναι γεγονός ότι η ιστορία αυτή ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια και τώρα μπορούμε να κάνουμε καλύτερες επιλογές. Αλλά να σας πω, δεν, το ζήτημα δεν είναι για τους 12 αυτούς τύπους. είναι για το ελάχιστο είδο, το, το, ελάχιστο αριθμό ιστοτόπων που μπορούν να μπουν ε, σε ένα εθνικό σύστημα και των οποίων το αποτέλεσμα spillover θα είναι τέτοιο ώστε να μπορέσει να έχει ε, ε, να αλλάξει ας πούμε το επιγραμμικό τοπίο της ε, χώρας. Είναι ένα είδος αργυρής σφαίρας κατά κάποιο τρόπο και με τον τρόπο αυτό θα, περάσουμε, θα ξεπεράσουμε και το πρόβλημα ε, της διαφοροποίησης. Δηλαδή όπου σε μερικές χώρες έχουμε μονάχα δημόσιες, ε, ε, δημόσιες δυνατότητες ενώ σε άλλες χώρες έχουμε συνδυασμό ιδιωτικών και δημοσίων. Δεν είναι μονάχα δηλαδή αυτά τα 12 είδη ιστοτόπων. Είναι η δυνατότητα διάχυσης του αποτελέσματος που θα έχουν στην, στη, τις ε, χώρες στις οποίες θα εισαχθούν και θα δημιουργηθεί με τον τρόπο αυτό και ένα, ε, μια καλή πλατφόρμα για τον ιδιωτικό τομέα από τον οποίο προκύπτουν οι θέσεις εργασίας, μιλισμονείτε. Όσον αφορά τώρα τα πρότυπα. Είχαμε τα πρότυπα ISO που δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβρη και ε, ε, βασιστήκαμε και στα ε, WACT βάσει του W3C που δεν είναι όμως ακριβώς πρότυπα. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι απολύτως ίδιες. Το θέμα λοιπόν του, των προτύπων είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι ένα δευτερεύον τεχνολογικό στοιχείο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε εναρμόνιση στα πλαίσια της οδηγίας. 8 Απριλίου θα έχουμε μια τεχνική συνεδρία η οποία θα συζητήσει εν λεπτομερία όλα αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Κοιτάξτε, ε, μπορούμε να συζητήσουμε διμερώς ε, όσον τώρα αφορά το θέμα της ε, τυποποίησης, αλλά να μην χάσουμε το χρόνο μας εδώ για αυτό. Βεβαίως το θέμα των τεχνικών προδιαγραφών δεν είναι τεράστιο με την έννοια ότι δεν υπάρχουν ατελείωτες δυνατότητες για τα κράτη-μέλη. Έχουμε ε, την περίπτωση των ευρωπαϊκών προτύπων και του ΆΙΖΟ ε, που ε, δεν κοστίζουν πάρα πολύ Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τα ευρωπαϊκά στάνταρ και τα ε, open standard. Οτιδήποτε μη ευρωπαϊκό θεωρείται open δηλαδή. Και θα πρέπει οι τεχνικές προδιαγραφές να είναι ίδιες έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Δεν είχα χρόνο να σας πω ότι εδώ και 12 χρόνια έχουμε χρησιμοποιήσει πολλά ε, χρήματα έρευνας, έχουμε χρησιμοποιήσει ήπια νομοθεσία, soft loss. έχουμε... Ε, έχουμε επιτύχει την συμφωνία των κρατών για τα ΟΑΚΑ του 2,0. Ε, Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν, μπορούμε, δεν είχαμε μπορέσει να επιτύχουμε τους εθνικούς στόχους γιατί δεν υπάρχει αντιστοιχεία της προσφοράς και της ζήτησης. Είδαμε ότι είχαν ε, τεθεί κάποιοι στόχοι για το 2010, ε, για το 2010 από χώρες οι οποίες δεν κατάφεραν τελικά ε, να επιτύχουν. Τώρα, οι δημόσιες ε, προμήθειες Κοιτάξτε, αυτό που προτείνουμε εμείς είναι να δούμε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυτά τα θέματα των εθνικών, ε, ε, των εθνικών αρχών, ε, από κάθε χώρα δηλαδή να υπάρχει ο expert, ο εμπειρογνώμονος ο οποίος ασχολείται με τα θέματα αυτά, να δούμε ακριβώς τι θέλουν και ε, έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι οποιοδήποτε αγοράσει κάτι είναι καλής ποιότητος ε, και δεν τροποποιείται από τη μια μέρα στην άλλη όπως γίνεται τώρα. Έτσι ώστε τα στάνταρ ναι μεν να είναι ίδια, αλλά δεν είναι εκεί το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ε, η επιθεώρηση, η εποπτεία, ο έλεγχος να είναι σωστός και να υπάρχει σαφήνεια, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, διότι η σαφήνεια δεν ήταν αρκετή. Σχετικά με την οριζόντια προσέγγιση εδώ του κ. Ταρκόφσκη, ναι, βεβαίω είναι ένα ζήτημα οι δημόσιε προμήθειες, αλλά πρέπει να ε, δούμε ότι οι περισσότεροι μεν ιστότοποι, οι εθνικοί δημόσιοι ιστότοποι ε, είναι αποτέλεσμα ε, δημόσιας προμήθειας, αλλά όχι όλοι. Και επίσης το σημαντικό δεν είναι πώς να δημιουργήσεις έναν ιστότοπο, το σημαντικό είναι πώς να τον λειτουργήσει και πώς η προσβασιμότητά του να διατηρείται στο χρόνο. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτείτε λίγο παραπάνω, think bigger λέει ο μιλητής. Να βρεθούν δηλαδή οι σωστοί τρόποι ε, να προχωρήσουν τα πράγματα και όσον αφορά τις ε, δημόσιες προμήθειες. Ε, τώρα, κατα εξουσιοδότηση πράξης, ξέρω ότι είναι κόκκινη γραμμή για τους περισσότερους. Εμείς θα αποσαφηνίσουμε σαφέστατα, έτσι ώστε να υπάρχει μεγάλη σαφήνεια για το ποιες και τι θα περιλαμβάνουν οι κατ' εξουσιοδότηση πράξης. Προσπαθούμε να το εξηγήσουμε στα κράτη-μέλη, δουλεύουμε μαζί τους να τους εξηγήσουμε τι κάνει ο καθένας και τι πρέπει να κάνει. Έχουμε δύο κατεξουσιοδότηση πράξεις, είναι σαφέστατο το γιατί ε, βρίσκονται εκεί. Θα το εξηγήσουμε όμως ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για το όσο μας ε, εξηγήσατε παντώντας. Πάρα πολύ ε, καλή αρχή θα κάνουμε για αυτή τη διαδρομή. Αλλά, όπως είπατε, θα τα ξαναπούμε, θα έχουμε και εκείνη τη μικρή υπήρξη. Θέλετε να ολοκληρώσετε και να μας πει και το χρονοδιάγραμμα. Χατζη Χατζημαρκάκης. Ναι, Πρόεδρε. Το κύριο θέμα είναι αν χρειάζεται η αξιολόγηση επιπτώσεων. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε εμεί να ισχυριστούμε ως κοινοβούλιο ότι δεν είναι απαραίτητο. Γι' αυτό λοιπόν ήταν και σημαντικό για μένα το να ακούσω τι έχουν να πούνε οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ για τις πολλές ε, υποδείξεις και εσείς κύριε Πρόεδρε Θέσε το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων. Τον είπατε ότι είναι πολύ ε, ε, παρεμβατική η προσέγγιση και πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο η λύση του soft law, του ενδοτικού δικαίου. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να πούμε, ε, και το λέω στην Επιτροπή εδώ, όπως άλλωστε το έχω πει και σε διμερείς σχέσεις, ότι είναι περίπλοκα αυτά τα οποία μας προτείνει. Δηλαδή τα πράγματα τα οποία καλούμαστε να προβάλλουμε σαν τυποποίηση είναι πολύ γραφειοκρατικά. Η υποχρέωση για κοινοποίηση, παραδείγματι. Πρέπει να φύγει, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχουν άλλοι σύγχρονοι τρόποι να επαληθευτεί εάν τηρεί ή όχι ένα κράτο μέλο την υποχρέωσή του. Και επίση, φρονώ ότι 12 χρήσει, εντάξει κύριε Τρασκόφσκι, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είναι περισσότερα ή λιγότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, με ένα μικρό αριθμό εφαρμογών να θεσπίσουμε το δίκαιο, όπως θα λέγαμε, με την δυνατότητα της πρόσβασης σε κάθε κράτος μέλος με ίσους όρους, γιατί είναι πολύ άνηση η μεταχείριση και πολύ ασαφής η κατάσταση. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα το περιλάβουμε και στο κείμενο. Βεβαίως ευχαριστώ πολύ για τα open standards που αναφέρατε. Εδώ είναι κάπως διαφυροποιημένη η πρόταση η ε, δική σχέση με τις επιτροπές, ε, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα, κύριε Έγκστρομ, να έχουμε ένα σαφές σύνολο προδιαγραφέων που θα εφαρμόζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδέα που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ και περιμένω την παρουσίαση και ε, της πρακτικής αργότερα. Κύριος Χάρμπουρ. Πρόεδρος. Οπότε θα το ξανασυζητήσουμε τον Απρίλιο. Για να δούμε. Για κάτω να βρω και εγώ το χρονοδιάγραμμα. Το σωστό. 25 Απριλίου και μετά το Μάιο ξανασυζητηθεί Ιούλιο ψηφορίας και Ολομέλεια τέλους Νοεμβρίου για ψηφορία. Να δούμε πώς θα πάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, κύριε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε καθυστερήσει Οπότε τώρα σκεφτείτε τον κύριο Μάντρε για μια παρουσίαση. Έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά αυτό το σημαντικό ζήτημα της συλλογική διαχείρισης δικαιωμάτων μεταξύ ιδιοκτησία και συγγενικών δικαιωμάτων εδαφική πολλαπλής ισχύω. Ε, επί τη ουσία έχουμε την κυρία Γκάλο, επίσης ε, η Ήτρε, έχει ασχοληθεί και άλλες επιτροπές είναι συναρμόδιες. Ο κύριος Μάντες ε, είναι ο συντάκτης. Άγκστρομ, Μακλάρκιν, είναι επίσης οι σκιώδες ηγητές. Ο κύριος Μάντες τώρα έχει το λόγο. Και έχουμε εδώ την τμήματάρχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα ε, της πνευματικής διοκτησίας και copyright. Μάντερς, ευχαριστώ. Πρόεδρε. Το χρονοδιάγραμμα το έχουμε συμφωνήσει με την κυρία Γκάλο. Οπότε ό,τι κάνουμε κι εμείς θα είναι σύντονο με το έργο της Νομικής Επιτροπής. Συνονεθήκαμε με τους και και όλοι συμφωνήσαμε ότι ε, έτσι θα προχωρήσουμε. Θέλουμε επομένως μεγαλύτερη διαφάνεια για καταναλωτές, για τους κατόχους των δικαιωμάτων και επίσης ε, προστασία και του δημιουργού. Σήμερα οι οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ε, ε, ίσπραξη των δικαιωμάτων, ε, είναι παντοδύναμοι οργανισμοί, παντοδύναμοι νομικά πρόσωπα και κάνουν μέχρι και 18 μήνες για να δώσουν τα χρήματα στους δημιουργούς. Και οπότε πληρώνονται αυτές οι εταιρείε, πληρώνονται αυτά τα νομικά πρόσωπα, αλλά χωρίς κανείς να ξέρει πώς γίνεται ο υπολογισμό, πότε θα πληρώσουν, πόσα θα πληρώσουν. Τέλος πάντων δεν είναι σαφές το πώς καθορίζονται τα σχετικά ποσά. Και επιγραμμικά και διασυνοριακά γίνονται αυτές οι συναλλαγές. Εν πάση πρέπει να έχουμε τελικά πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Εάν κάποιος είναι πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικά, τότε θα πρέπει να καταβληθούν τα σχετικά χρήματα σε αυτόν τον πάροχο. Εγώ λέω να θεσπίσουμε και εδώ μια μόνο απευθυντική θηρίδα. Κάπως συγκρίνεται η κατάσταση εδώ με την συλλογή, με την ίσπραξη των φόρων. Όμως για τους φόρους είναι ξεκάθαρο πόσα και πού πρέπει να καταβληθούν ως φόρος. Δεν θέλω να έχουμε πολλαπλασιασμό των γραφειοκρατικών κρατικών οργανισμών, όμως θα πρέπει να υπάρχει κάποιος φορέας διαχείρισης αυτών των δικαιωμάτων. Και να υπάρχει επομένως κάποιο είδους ε, τιμολόγιο που να καθορίζεται με σαφήνεια το πόσα οφείλονται. Και θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία αυτών των νομικών προσώπων συλλογικής διαχείρισης. Να υπάρχει βεβαίως και σχετική προθεσμία για αυτό το τιμολόγιο. και επίσης να είναι σαφές το πότε τελικά ο εισπράξας οργανισμός θα καταβάλει στον ε, δημιουργό. Και δεν τους λείπουν τα χρήματα καθόλου αυτών των οργανισμών. Τα επενδύουν αντί να τα δώσουν στον δημιουργό, στον καλλιτέχνη. Και φυσικά θα πρέπει να αποτρέψουμε αυτούς τους οργανισμούς να επενδύουν τα χρήματα σε επικίνδυνες τοποθετήσεις. Να ενεργήσουμε δηλαδή προς το συμφέρον των καλλιτεχνών. Επίση, δεν θα πρέπει να υπάρχει δεσμενή διάκριση σε σχέση με το από πού προέρχεται ε, ο κάθε τέτοιο εισπρακτικό ε, οργανισμό. Τελικά ο καταναλωτή επομένω καταβάλει αυτά τα πνευματικά δικαιώματα, όμω θα πρέπει να χαρακτηρίζεται αυτό το καθεστώ από διαφάνεια. Κάτι το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Γι' αυτό και έχουμε μεγάλε διαφορέ από τόπο σε τόπο. Όποτε γεννώνται πάντως διαφορές, δεν θα πρέπει να γίνεται δικαστική επίλυση τους γιατί σε αυτή την περίπτωση και οι δύο διάδικοι έχουν να πληρώσουν πάρα πολλά δικαστικά έξοδα. Και εγώ δικηγόρος είμαι και τα ξέρω. Καλό είναι να υπάρχει δουλειά αλλά όχι όταν, όταν υπάρχει άλλη λύση. Να υπάρχει λοιπόν, κάποιο είδους επιδιαιτησία, κάποιο είδου συμβιβασμό να βρεθεί κάποιος τρόπος να γίνεται εξώδικος σε συμβασμός ας πούμε. Και έτσι επομένως να ρυθμίζονται διαφορές μεταξύ καλλιτεχνών, δημιουργών και αυτών των εισπρακτικών ε, νομικών προσώπων. Στι 25 Απριλίου, επομένω, θα σα υποβάλω την έκθεσή μου. Περιμένω πώ και πώ να πούνε τη γνώμη του συνάδελφοι, να μου πούνε σε ποια σημεία συμφωνούν και να δούμε ε, τελικά σε ποιο σημείο θα επιτευχθεί η συμφωνία. σω είναι δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Good, thank you. Uh, thank you very much, Well, Αντουάν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα ήρθε η σειρά των ε, σχεδόν εισηγητών για να δούμε ποιο είναι στην Α, η κυρία Γκέμπου Έχετε το λόγο. Ναι, ναι, ναι μπορεί να πει Sorry, it's, yeah. Sabine, okay. sorry. Yeah. Ε, no problem at all. Ε, Κυρία Φερχέλιεν, ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την παρουσίαση των ιδεών του κύριου Μάντερς. Εγώ Όπω είπα και στην συνεδρία των Σκιωδών, δεν είμαι πεπισμένη τελείω για αυτή την ιδέα του one-stop shop, τη μονοθεριδικής προσέγγιση. Δηλαδή να μπουν τα πάντα μέσα στο ίδιο, ε, στην ίδια αρχή που θα γίνει μια υπεραρχή θα λέγαμε. Δηλαδή κάθε είδους ε, λογαριασμός, διαμεσολάβησης, δικαιώματα θα μπουν όλα στο ίδιο σημείο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Υποστηρίζω όμως την ιδέα ότι πρέπει κάτι να γίνει διαχρονικά που θα είναι και ε, αξιοποιήσιμο για τον χρήστη της ε, άδεια για οποιονδήποτε θέλει να κατεβάσει μουσική από το διαδίκτυο, να χρησιμοποιήσει τη μουσική, ε, να παίξει τη μουσική αυτή στο καταστημά του που θέλει να αξιοποιήσει για δική του παραγωγή ενδεχομένω ένα μουσικό κομμάτι. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να είναι δυνατόν να τα συναντά σε ένα σημείο σχετικά οργανωμένο μέσα στο διαδίκτυο για να υπάρχει η σχετική δυνατότητα για την ε, ε, συνεννόηση και τα τέλη. Έτσι λοιπόν, να υπάρχει μια βάση δεδομένων όπου όλα τα δικαιώματα και οι άδειε να συναντιούνται και να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να πάει να ρωτήσει, να πάρει πληροφορίες ή άδεια για μια μορφή χρήσεω, χωρίς όμως απαραίτητα να είναι το ίδιο σημείο, με τον ίδιο τρόπο για τους πάντες. Δεν θέλω μια νέα αρχή δηλαδή ή ένα νέο οργανισμό. Θα ήταν υπερβολικό αυτό. Και δεν, χρειά... βοηθάει και στη διαφάνεια. Ξεκάθαρα πρέπει, πιστεύω, και ίσως το λέω επειδή είμαι και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού ταυτόχρονα, η, ε, υπηρεσίες αξιοποίησης να μην περιορίζεται μόνο στην οικονομική διάσταση αλλά και στην πολιτιστική. Μια εγγύηση λοιπόν, μια διασφάλιση της πολιτισμικής πολυμορφίας, ποικιλία είναι και το να έχει την προστασία αυτήν ο μικρός παραγωγός, ο όχι γνωστός, να μην είναι μόνο η μεγάλη εταιρεία δίσκων αυτή που θα μπορεί να προσφέρει το υλικό της, αλλά και η λιγότερο γνωστή. Οι δομές ε, στον χώρο του, της, των οπτικοακουστικών μέσων δεν μπορούν να αντιγραφούν ε, μία προς μία. Υπάρχουν διαφορετικές δομές ε, και όσο και αν θέλουμε δεν μπορούμε να τις ε, επαναλάβουμε όπως έχουμε, να τις μιμηθούμε. Και νομίζω ότι οι διασυνοριακές άδειες δεν καλύπτονται επαρκώς στην πρόταση. Χρειαζόμαστε δομές οι οποίες να επιτρέπουν τη συνεργασία πέραν των συνόρων και μια δυνατότητα διαμεσολάβηση ενδεχομένως όταν έχουμε διαφορετικούς κατόχους δικαιωμάτων, δικαιούχους δηλαδή, ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να ε, ξεκαθαρίσει με μια υπηρεσία αξιολόγησης, αξιοποίησης ποιος ε, είναι ο δικαιούχος στον οποίο θα πρέπει να αποτανθεί στην κάθε περίπτωση. Και επίσης μεταξύ Αυτόν και του χρήστη, θα πρέπει να δούμε εάν μεγαλύτερη σημασία έχει ο χρήστης, ο οποίος ενδεχομένω παίρνει ένα playlist, μια λίστα μουσικής, ε, μπορεί να έχει ταχύτερη πρόσβαση ή αν πρέπει να ε, ψάχνει ένα τα κομμάτια της μουσικής που τον ενδιαφέρουν. και να τα μεταφέρει σε μια δικιά του λίστα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και την πρακτική διάσταση. Yeah, αξιοποίηση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο βελτιωμένο και στην ε, πλειοδοσία να υπάρχει χρόνος ε, για αντίδραση. Γιατί πρέπει να είναι σε θέση και ο χρήστης να γνωρίζει πού, πώς, με ποιους όρους για την Γενική Συνέλευση στα, στην ε, ε, διαδικασία αυτή της αξιοποίησης των πνευματικών ε, δικαιωμάτων, η εταιρεία, την εταιρεία διαχείρισης δηλαδή, μπορούμε να έχουμε μία συλλογική διαχείριση με ένα, αλλά τελικά ο ίδιος ο πνευματικός δημιουργός είναι ο παράγον, το σημαντικό στοιχείο αυτής της εταιρείας διαχείρισης. Και μην ξεχνάμε ότι αν ε, επιβάλλουμε πολλές διατυπώσεις ε, θα καθυστερήσει, θα επιβραδενθεί, θα ε, δυσκολέψει το έργο της εταιρείας διαχείρισης. Δεν πρέπει δηλαδή να επιβάλλουμε υπερβολικές διατυπώσεις. Και θα πρέπει να αναλογιστούμε πολύ προσεκτικά πού θα είναι πιο λεπτομερείς οι διατάξεις και πού λιγότερο. στο άρθρο 33, το οποίο επίση θεωρώ σημαντικό, έχουμε την ε, δυνατότητα της, του διαδικτυακού προγράμματος από το ραδιόφωνο. και εκεί δεν έχω αντίρρηση. Ως προς την χρήση της οδηγίας ε, παροχής υπηρεσιών και στην εταιρεία διαχείρισης, δεν είμαι βέβαιη ότι είναι τόσο εύστοχη αυτή η λύση. Γιατί έχουμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα βάθους και εύρους διατάξεων και διατυπώσεων σε κάθε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Και έτσι μπορεί κάποια κράτη-μέλη να έχουν μία πολύ αυστηρή και παρεμβατική, επεμβατική καλύτερα, νομοθεσία, ενώ κάποια άλλη κάποια άλλη να έχουν πολύ πιο χαλαρές διατάξεις. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή ότι μπορούν τα πάντα να ταυτιστούν, να βρούμε ε, ομοιότητες παντού. Στο 10.2 δεν είναι σαφή η διατύπωση. Η επιχείρηση, η εταιρεία διαχείρισης είναι λίγο πολύ καταπιστευματοδόχος, δεν έχει στην ιδιοκτησία της αυτά τα δικαιώματα και πρέπει να οριστεί ένα χρονικό σημείο μέχρι το οποίο πρέπει να έχουν καταβληθεί τα ποσά. Γιατί φαντάζομαι ότι κάποιοι πληρώνουν εγκαίρως, κάποιοι πιο αργά. Αυτό κάπως πρέπει να προσδιοριστεί. Διαφάνεια, σαφής όροι και διατάξεις είναι για να ολοκληρώσω το πιο σημαντικό από όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι για τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσατε το θέμα δείχνει την περιπλοκότητα του θέματο, αυτού, κυρία Γκέπχαρτ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Βάιντεν Χόλτσερ με παρακάλεσε να τον εκπροσωπήσω εδώ. Λόγω των απεργιών που είχαν αναγγελθεί από τη Λουφτχάνσα, από τον προσωπικό τη Λουφτχάνσα, επέστρεψε χθε στην ε, έδρα του και έτσι δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα. Με παρακάλεσε να τον εκπροσωπήσω, αλλά δεσμεύεται ότι από εδώ και μπρος θα είναι πάντοτε παρόν σε συζήτηση το θέμα αυτό. Πάντως ευχαριστώ πολύ για την ε, συνεργασία, τον κύριο Μάντερς. Θεωρεί ότι πάντα υπάρχει περιθώριο καλή συνεργασία, αν και πάντα υπάρχουν κάποια σημεία που θα μπορούσε κανείς να ξαναμελετήσει, όπως αυτό της ενιαίας συμμονοφυριδικής ε, προσέγγισης και εδώ δεν έχω εγώ δική μου θέση να... δεν έχω εδώ δικές του υποδείξεις, δική μου θέση προβλέπω, ε, παρουσιάζω. Η λύση λοιπόν εδώ είναι πολύ σημαντική για την ψηφιακή εσωτερική αγορά, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο προτείνεται, αλλά ο, ο θεωρεί ότι πρέπει για την εταιρεία διαχείρισης των δικαιωμάτων να ε, φροντίσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αδιαφάνειας του τρόπου με τον οποίο εργάζονται οι εταιρείε διαχείρισης, τον τρόπο τον οποίο εργάζονται οι εταιρείε διαχείρισης. Πρέπει να δούμε πόσο υπολογίζονται τα τέλη, τα δικαιώματα, ποιος θα υπολογίζει, με ποιο χρονικό ορίζοντα και γιατί γιατί μπορεί για κάποιον καλλιτέχνη να παρουσιαστεί ακόμα και τρία, παρουσιαστεί ακόμη και καθυστέρηση τριών ή τεσσάρων ετών. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι, με κάτι πρέπει να βιοποριστούν. Δεν είναι όλοι εκατομμυριούχοι όπως ε, ίσως κάποιοι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, πολύ γνωστοί. Πολλοί είναι απλοί βιοποριστές που ζουν με τα ελάχιστα. Και έτσι πρέπει και αυτούς να τους λάβουμε υπόψη. Έτσι λοιπόν, αυτά τα πολύ περίπλοκα συστήματα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να τα δουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι δύσκολο να τα κατανοήσουν και γι' αυτό καλό θα ήταν να έχουμε μία κοινή ε, ένα κοινό σύνολο κανόνων, ε, παραδείγματι για την ε, διασυνοριακή αδειοδότηση και κυρίως αν πρόκειται για την ε, πολλαπλή αδειοδότηση που αυτή τη στιγμή απαγορεύεται ή άλλα στοιχεία, άλλες λεπτομέρειες που θα πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά. Επίσης, στη γνωμοδότηση της ΣΥΜΚΟ, σημείο 1 και 2, η όροι πρόσβασης και η διαφορά μεταξύ της ε, ε, πρόσβασης και του προϊόντος, του πολιτιστικού υλικού. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές άδειε πέραν των συμβατικών που γνωρίζουμε, όπως τα Creative Commons, λύσεις τις οποίες ε, δεν είναι πάντα σε θέση να αξιοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες γιατί είναι δεσμευμένοι σε συμβάσεις, σε συμβόλαια που τους περιορίζουν ως προς την αναζήτηση άλλων λύσεων. Πρέπει λοιπόν να δούμε και αν υπάρχουν δυνατότητες να διευκρινίσουμε αυτή τη διάσταση. Δεν θα σας διαβάσω όλη την επιστολή του συναδέλφου, αλλά πάντως θα ήθελα να πω ότι η διαφάνεια, η ε, αντιμετώπιση των δεσμευτικών όρων, η εναλλακτική διευθέτηση διαφορών, και εδώ έχουμε προχωρήσει σημαντικά ως προς, τον, προς τη ρύθμιση. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα βήματα πρόοδου. Οι άδειε που δεν είναι σαφείς ως προς την αδειοδότηση της χρήσεως σε οπτικο-εκουστικές υπηρεσίες ή σε ε, μουσικά ρεπερτόρια. Όλα αυτά πρέπει να ε, συζητηθούν. Επίσης θέλουμε μεγαλύτερη και ευρύτερη προσφορά μέσων, προσαρμογή των συστημάτων αδειοδότησης στην δικτυακή εποχή, ε, περισσότερες ε, δυνατότητες ανταγωνισμού και στις εταιρείες διαχείρισης, διαφάνειας εταιρείες διαχείρισης και άλλα τέτοια ζητήματα που έχει επισημάνει ο συνάδελφος και που πιστεύω καταδεικνύουν την πληθώρα των προβλημάτων και ταυτόχρονα τη σημασία του ζητήματος για όλους μας. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ για μία ακόμα φορά. Ευχαριστώ στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είχαμε μια δημόσια ακρόαση αυτή τη βδομάδα ε, σχετικά με την ε, έκθεση αυτή και μάλιστα, την, ε, και μάλιστα Η αίσθηση που έχω από την Νομική Επιτροπή είναι ότι συμφωνεί με στα ουσιώδη πράγματα και εδώ ακούγοντας τους παριστάμενους έχω την ίδια αίσθηση και επομένως αυτό μου δίνει ελπίδα ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, με κάποια μεγάλη πλειοψηφία επί κάποιων ε, σημαντικών στοιχείων. Για μένα το σημαντικότερο θέμα πέραν αυτών που ανέφερε και η κυρία Γκέπχαρτ, είναι ότι τα χρήματα δεν πληρώνονται έγκαιρα και με τον κατάλληλο το σωστό τρόπο. Στην ε, μελέτη αντικτύπου του Κομισιόν αναφέρεται ότι 5,7 δις και το τονίζω δις ευρώ έχουν συλλεγεί από τις ε, υπηρεσίες ε, ε, συλλογικής διαχείρισης χωρίς να τα έχουν αποδώσει όμως τα χρήματα αυτά. Δεν ανήκουν στις εταιρείε, ανήκουν στους συγγραφείς ή στους συνθέτες. Επομένως χρειάζομαστε μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη λογοδοσία και φυσικά τους σωστούς κανόνες οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι τα χρήματα πληρώνονται σωστά με ενδιαφέρει πολύ το άρθρο 2 παράγραφος 2, συγγνώμη, το άρθρο 12 παράγραφος 2. Ότι δηλαδή αν για πέντε χρόνια δεν βρεθεί ε, ο δικαιούχος, τότε οι υπηρεσίες συλλογική διαχείριση έχουν δυνατότητα να κρατήσουν τα χρήματα. Ε, νομίζω ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε. δεν είναι δυνατόν ε, να επιβραβεύονται εν τέλει οι υπεύθυνοι των εταιριών αυτών επειδή δεν προσπάθησαν και δεν κατάφεραν να βρουν ε, τον ε, δικαιούχο. Κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να βρει τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής των αποφάσεων στην χώρα. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι αποφασίσαμε ότι ε, οι βιβλιοθήκες ας πούμε πρέπει να πληρώνουν αποζημίωση δικαιούχος ε, για τα ηλεκτρονικά βιβλία τα οποία ε, διαθέτουν. Επίσης, Ε, εν πάση περιπτώσει όμως ε, τα, ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν για τις λεπτομέρειες αλλά το βέβαιο είναι, είναι ότι δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε ε, τους, τις υπηρεσίες συλλογής χρημάτων ας πούμε να και εισφορών ε, να κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως είπα και προηγουμένως και εδώ θα σταματήσω και με αυτό θα σταματήσω, είναι ότι ε, έχω την αίσθηση ότι στην Επιτροπή διαφαίνεται μια συμφωνία και επομένως ότι θα μπορέσει τελικά να συμφωνήσει επί των κεντρικών ε, γενικών γραμμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και είναι καλό που δουλεύει για τα θέματα ιστορικής αγοράς στην Νομική Επιτροπή θέλει κανείς άλλος να μιλήσει, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο, σας λέω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ ε, με την ε, ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε και να βελτιωθούν τα δικαιώματα των καλλιτεχνών και να, έχουν, να βρεθούν υπό έλεγχο οι εταιρείε οι οποίες κάνουν την συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Αυτό είναι θέμα εσωτερικής αγοράς είναι παθιασμένος ο κύριος Μάντερς και έχει επιδείξει μεγάλη ευρηματικότητα σε πολλά σημεία της εκθεσής τους. Αλλά δυστυχώς αυτό το one-stop shop, η μονοπευθυντική θηρίδα δεν με βρίσκει σύμφωνη. Ε, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως εμάς μας απασχολεί η αλλω μα μας πρόθεση αυτών των, ε, ε, των δικαιωμάτων και νομίζω ότι αυτή η μονοπευθυντική θηρίδα δεν μπορεί να βοηθήσει ε, ιδιαίτερα. Εν πάση περιπτώσει το ζήτημα είναι πόσο μπορούμε να επιτρέψουμε περισσότερες εδαφικές ε, ε, αδειοδοτήσεις και πόσο μπορεί να προωθηθεί η διασύνδεση αυτών των μονάδων. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ελεγχθούν οι διαδικασίες οι οποίες ήδη υφίστανται για να δούμε ότι λειτουργούν σωστά και έχουν ληφθεί ε, τα απαραίτητα μέτρα. και ε, εν πάση περιπτώσει όποια απόφαση και να πάρουμε θα πρέπει να είναι σωστή απόψη κόστους ωφέλους, από την απόψη σχέση κόστους ωφέλους. Θα αναφερθώ τώρα σε κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως σαφής. Ε, πρώτα απ' όλα σαφής ορισμός των ε, εταιριών συλλογικής διαχείρισης που βρίσκεται στο άρθρο 3. Νομίζω ότι ε, δυνάμει του άρθρου αυτού μπορεί να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνη. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, εάν δεν έχουμε σωστή εφαρμογή του πεδίου, ε, να ε, δημιουργηθεί ένα playing field το οποίο θα είναι ίδιο για όλους. Επίσης, αναφέρεται ότι εάν για πέντε χρόνια δεν έχει βρεθεί ο δικαιούχος από πλευρά της εταιρεία λογικής διαχείρισης, τότε αυτή μπορεί να κρατήσει τα δικαιώματα νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις, να πούμε ενδεχομένως ότι τα χρήματα αυτά δεν τα κρατούν, αλλά ε, μπορούν να τα επενδύσουν με συγκεκριμένους τρόπους κτλ. Ε, επίσης ότι τα χρήματα θα πρέπει να δίνονται συχνά ε, και με σωστό τρόπο. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να εκλειφθεί ως μία ε, κατά ε, τακτά διαστήματα καταβολή των χρημάτων έτσι ώστε ε, να διασφαλίζεται και μια καλή ροή εισοδημάτων για τους ανθρώπους αυτούς. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τους και Η κυρία Πάτστρα, μήπως θα μπορούσε να, να απαντήσει ένα-δυο λεφτάκια στα πιο σημαντικά. Έχουμε ψηφοφορίες να κάνουμε, οπότε παρακαλούμε να είστε σύντομοι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομοι και ξεκινώ αναφέροντα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεγάλη τη Χαρά επανέρχεται εδώ στην ΙΜΚΟ για να συζητήσουμε αυτή τη φορά την ε, οδηγία για τη συλλογική διαχείριση. Και ε, άκουσα όλου όσου το λόγο και κατά τη γνώμη μας ε, είναι ποιοτική η συνεργασία με το Κοινοβούλιο και πάρα πολύ σημαντική γιατί εδώ και πολύ καιρό θέλατε να υπάρχει μια τέτοια οδηγία από τις τραπέζες οπότε να και τελικά εμείς την κατεβάσαμε την, την πρότασή μας και ε, μιλούμε για πάλι πολύ εντατική δουλειά με, με πολλές ώρες και ξέρετε περισσότερο είμαι στο Κοινοβούλιο από ό,τι στο γραφείο μου για, για αυτή την υπόθεση το οποίο δεν πειράζει βέβαια Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους προτείνουμε αυτή την οδηγία ήδη ε, αναφέρθηκαν από όσο το λόγο και από τη μία μεριά έχουμε την προβληματικό τρόπο ή ε, από κάποια τέτοια νομικά πρόσωπα όσον αφορά το τι κάνουν τα χρήματα, δεν υπάρχει διαφάνεια σε όλη αυτή τη διαχείριση κλπ. Αλλά έχουμε και, και άλλα προβλήματα κατά τελευταία δεκαετία, το ότι στην ψηφιακή ενιαία αγορά υπάρχουν νέα προβλήματα. Έχουμε επίσης και για αυτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες επιγραμμικά αδειοδοτήσεις που αφορούν πάνω από μία χώρα. Επομένως γι' αυτό προσπαθήσαμε να δώσουμε μία αντίστοιχη δομή για διάρθρωση σε αυτή την οδηγία. Θέλουμε να καλύψουμε όλες αυτές τις ε, εταιρείε συλλογικής διαχείρισης. Επίσης ε, προσπαθούμε να ασχοληθούμε, να θίξουμε και τα επιγραμμικά προβλήματα. Επίσης ε, να καλύψουμε και τις περιπτώσεις δικαιωμάτων που αφορούν έργα μουσικής περιπτώσεις που έχουμε δημιουργία οπτικοακουστική, επίσης όταν έχουμε αδειοδοτήσεις που αφορούν πάνω από μια χώρα και έχουμε από μια μεριά τα δικαιώματα των ε, παραγωγών ή των ε, εκτελεστών. Εκεί δεν υπάρχει σωστή διαχείριση. Συνήθω η παραγωγή δεν τι εγκρίσει και τι άδειε αναπαραγωγή κλπ. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό και δεν φύγουμε αυτό ακριβώς ε, όμως η μουσική καλύπτεται όσον αφορά τα οπτικοακουστικά. Πώς κανείς λοιπόν θα παράσχει ε, download, δηλαδή δυνατότητα να κατεβάσει κανεί από το ίντερνετ κάποιο τέτοιο οπτικό ακουστικό δημιούργημα, οπότε τότε χρειάζεται να προβλέπεται η σχετική αδειοδότηση και η σχετική ρύθμιση. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του να καλύψουν αυτές τις λεπτομέρειες για ε, να καλύψουν ότι έχουμε σε κάθε κράτος μέλος διαφορετικά είδη ε, τέτοιων εταιρεών διαχείρισης, υπάρχουν διαφορετικές ε, εταιρείε, διαφορετική παράδοση σε κάθε χώρα γιατί πολλές φορές πρέπει να καλυφθούν διαφορετικά είδη ε, συμφωνιών και αμοιβών. Πάντως, για να επαναλάβω αυτό το πηγαν πολύ, θα πρέπει να καλύψουμε την ψηφιακή ενιαγορά, τις ε, διασυνοριακές εγκρίσεις, ε, πάρα πολλές ε, από αυτές τις εταιρείες δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις καινούργιες ε, μορφές. Χρειάζεται κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές δυνατότητες και γι' αυτό θα πρέπει και να καλύψουμε τις πολιτιστικές διαφορές στην πολιτιστική πολυμορφία. Να μην σας πάρω άλλο από το χρόνο. Μεγάλη μας χαρά τα είπαμε και θα ξανασυζητήσουμε για να συζητήσουμε και για τη μορβευτική θηρίδα, αλλά και αυτό μας απασχολεί. Δεν θέλουμε να έχουμε επιπλέον γραφειοκρατία. Πάντως, πάντως, ευχαρίστως με τους ε, συνεισηγητές να συζητήσουμε τις ιδέες τους. Εμείς, ευχαριστούμε, λέει ο με μεγάλη μας χαρά, πάντοτε σας υποδεχόμεθα εδώ στην Ήμικο. Τώρα, κύριε Μάντρες, έχω τώρα το χρονοδιάγραμμα πρέπει να μα τα πείτε κι εσείς, αν θέλετε να συνοψίσετε, να δευτερολογήσετε, να κλείσουμε, για να πάμε για την πληροφορία. Μάντερ. Έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί όλοι μιλούν για όρους θεμητού ανταγωνισμού, αλλά εγώ θέλω να ε, έχω ένα φορές διαχείριση, το οποίο δεν είναι ανταγωνισμός αφού είναι μόνο ένας. Τέλος πάντων, ε, θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα τη μετάφραση, θα πρέπει να το μελετήσουμε στις 25 Τετάρτου εδώ, θα συζητήσουμε 14 Πέμπτου τροπολογίες, η προθεσμία, ψήφιση στην Επιτροπή 8 ε, Έκτου και 9 Εβδόμου στην Γιούρη. Ψηφοφορία δηλαδή στην Επιτροπή. Ο πρόεδρο εκτός μικροφώνου. I'm Sorry we've run over a bit, but I think it was definitely uh, worth uh, completing that item. Uh, when... Έχουμε μείνει πίσω με το χρονοδιάγραμμα μας, αλλά όμως ήταν αξίζει, είναι ενδιαφέρον το θέμα και τώρα πάμε να ψηφίσουμε. Κλινικές δοκιμές φαρμάκων. Αυτό το έχουμε συζητήσει και έχουμε ε, χθες που συζητήσαμε, συζητήσαμε αυτές τις τροπολογίες. Γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, κοιτάξτε αν έχετε μαζί τις κάρτες. Όσοι ψηφίσετε Don't tell me. I've erroneously picked out my Tesco club card. Την ξεχάσετε εσείς. Αχ, ναι, ναι, για πήρα του το σούπερ μάρκετ. Πήρα του Tesco την κάρτα αντί για την κάρτα ψηφοφορίας. Συμπαθάτε με. Δεν την έχω, δεν την έχω, λέει κυρία Πρέντεργας. Just keep an eye on you over here then. Yeah, sorry about that. Okay, right. Uh, so is everybody ready? Well, we have. But uh, Anna is coming. All right.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 Όχι, όχι, όχι, να, να κάνουμε κατευθείαν ε, ε, ηλεκτρονικό έλεγχο. So, has everybody got their cards in? Έχετε βάλει όλοι τις κάρτες στο μηχάνημα, κύριε Πέντερκα, το ξέχασε, είναι κατά, πέρα της εφορίας. 23, 10. 61. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί είναι οριακό το αποτέλεσμα. 20-14 γίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 64 έχει αποσυρθεί. 65. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Έλεγχος για το 68. Ψηφίζουμε. 16-18 απορρίπτεται. 69. Βερνιό. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 71 ε, με προφορική τροπολογία ζουγά, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 72, Μακλάρκιν, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική, αριθμόν 1, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 75 και 76, υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 77, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 78, υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος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 Έλεγχος. 79. Πέρας. And that's rejected. Απορρίπτεται. 17-17. 80. Υπέρ. Κατά. Ογδόντα 81. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Those in favor. Those against. That's... Υπέρ κατά και επομένως με το ζόρι περνάει. 82. Those in... 82. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 83. 84 υπέρ κατά απορρίπτεται 85 υπέρ κατά και αυτή απορρίπτεται 86 υπέρ κατά απορρίπτεται 87 υπέρ κατά απορρίπτεται 90 υπέρ κατά και αυτή απορρίπτεται 91 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 7. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται έλεγχος ηλεκτρονικός για την 100. Εκατόν ένα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. δύο Υπέρ. Κατά. Και αυτή είναι εγκρίνεται. 103. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 104. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίσουμε τις ε, τροπολογίες Μακλάργιν όλες μαζί με τις προφορικές τροπολογίες και αυτές τις τροπολογίες παραγράφους, όλες αυτές μαζί που βλέπετε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Όλες μαζί εγκρίνονται. 113 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 117 του εισηγητού κυρίου Ζουβέν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τρία, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. είκοσι, υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφορία για το εκατόν, είκοσι. Απορρίπτεται μια που είναι 17-17, ισοψηφία. Α, όχι δεν είναι, 18-17. Άρα δεν είναι ισοψήφια. 110, μπουσόι. Συμβαστική 4, συγγνώμη πριν ήταν η 10. Ε, συμβαστική 4, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 118, μπουσόι, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 123 ζωέ, 124 βελή. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 128 ρίλε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 130 ζουβάν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 121. Υπέρ για το 121. Κατά. Εγκρίνεται. 110. Υπέρ. Έλεγχος για το 110. Ψηφίζουμε. Πέραση ενέα 9 και 12 από κοινού υπέρ. Κατά εγκρίνονται. 13. υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 132 υπέρ. Κατά εγκρίνονται. 130 3 με την προφορική τροπολογία που τη βλέπετε εκεί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 με τις προφορικές τροπολογίες του κ. Μπουσό και μια αιτιολογική παράγραφος υπέρ, κατά, εγκρίνεται 142 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 143 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 144 145 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 146 και 148 από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 147 υπέρ, κατά. Τι λένε οι φιλελεύθεροι, α, είστε υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 150 υπέρ. Έλεγχο για το 150. 150 πέρα ψηφορίες απορρίπτεται. 17, 18, 151 Χωριστή ψηφοφορία υπέρ για το πρώτο τμήμα, κατά. Εγκρίνεται το πρώτο, δεύτερο, υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα, 152, υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154, υπέρ κατά 154 έλεγχος ψηφορίας εγκρίνεται 16-14 156 ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ. Έλεγχος 158. Πέρασε της εφορίας. 20 20-14 εγκρίνεται. 159 που είναι συμβατή. 159. Πέρασε ο απορρίπτεται με 15-18. 60 υπέρ. Κατά αποχές 161. Ποιοι είναι υπέρ. Πρέπει να κάνουμε έλεγχο για το 161. 2014. υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 167 υπέρ κατά. 167 έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 14-18. 168. Υπέρ. Κατά. Το 68 ψηφίζουν. πέρας Απορρίπτεται. 17-17. 169 υπέρ. Ψηφίζουμε για το 169. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. 171. Ε, έλεγχος για το 171. Πέρας. 13-20 απορρίπτονται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 174. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 175. Υπέρ, κατά. Κατά 76. Υπέρ, κατά. Έλεγχος για το 176. Πέρασε. 20-14. 178 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά, εγκρίνεται, 21, εγκρίνεται, 180, χωριστή ψηφοφορία, υπέρ, κατά, το πρώτο τμήμα εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, υπέρ, δεύτερο τμήμα, ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ έλεγχος για το 182 Πέρα τη εφορίες εγκρίνεται 183 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 185 υπέρ. Έλεγχος. 185. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά. χέρι συγκρίνεται 24 υπέρ. Κατά. χέρι εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 190 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 196. Έλεγχος για το 116 λέει ο πρόεδρος τώρα. 116. Πέρασε. Δεκαέξι δεκαεπτά. Απορρίπτεται. 195. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 196. Συγγνώμη, λέω ο πρόεδρος, 26. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 196. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 197. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 198 υπέρ κατά εγκρίνεται. 199 υπέρ κατά εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά εγκρίνεται. 200 υπέρ κατά εγκρίνεται. 201. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ιτιολογικές παράγραφοι. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 44 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155 κατά 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά έλεγχος ηλεκτρονικός για το 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 54, υπέρ, κατά, αποχές, άρα κάνουμε ηλεκτρονικό για το 54, ψηφίζουμε. Πέρας, 19, 14, 55. Μακλάρκιν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επομένως τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε το σύνολο της προτάσεως της τελικής. Ψηφίζουμε. Πέρας. Κατά κύριε Πρέντεγκαστ. Εγκρίνεται 19-14. Χωρίς αποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπουσό για το έργο που επιτελέσατε και θα συνεχίσετε στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πριν αποχωρήσετε, θα ήθελα να σας ζητήσω να προβούμε σε επίσημη έγκριση με ψηφοφορία του νέου χρονοδιαγράμματος για τις ε, συνόδους. Γιατί έχουμε τη, τη, μία κατάσταση με την έξτρα ολομέλεια. Εγκρίνεται, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ αυτούς που ήρθαν να ψηφίσουν. Και τώρα θα κάνουμε την έκθεση της κυρίας Γκέμπχαρτ. Θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Έχουμε, Έχουμε καθυστερήσει, αλλά θα πάμε λίγο πιο γρήγορα τώρα. Να παρακαλέσω όσους σκοπεύουν να αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν χωρίς φασαρία για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Κυρία Γκέμπχαρτ. Έχετε το λόγο για να κάνετε την παρουσίαση της γνωμοδότησης και των τροπολογιών σας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. 51 οι τροπολογίες, τις οποίες βρίσκω εν γέννη επικοδομητικές, θετικές. Μπορούμε, πιστεύω, χάρη σε αυτές να κάνουμε μια καλή γνωμοδότηση για την ε, δυνατότητα με τη βιομηχανική πολιτική να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα της Ευρώπης. Είναι καλό πιστεύω, όπως είχα πει και την άλλη φορά, να συζητούμε τη βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη πλέον, γιατί η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, η οικονομική κρίση, είναι νομίζω ε, και ένας τρόπος να διαπιστώσουμε ότι χρειαζόμαστε όχι μόνο υπηρεσίες αλλά και βιομηχανία. Εάν ο ένας κλάδος αντιμετωπίζει προβλήματα, τουλάχιστον μπορεί να λειτουργεί καλύτερα ο άλλος κλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πρέπει σήμερα. Είναι θετικό επίσης το ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών αναλαμβάνει ένα μέρος αυτής της εργασίας, γιατί έχουμε να κάνουμε όντως με την εσωτερική αγορά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξελίξη όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική είναι, όπως ξέρουμε, πολύ διαφορετικές και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα περάσω τώρα λίγο εν τάχει τις τροπολογίες ε, για να πω κάποιες ε, απόψεις. Καταρχάς ξεκινώ με τον κύριο Χατζημαρκάκη θα αναφέρουμε τους, ε, ανάλογα με τον συντάκτη της τροπολογίας. Είναι πολύ επικοδομητικές οι τροπολογίες του, με βοηθούν διατέρος και τον ευχαριστώ. Ιδιαίτερα η παριθμόν 4 εντάσσεται ακριβώς στη γραμμή αυτή την οποία σας περιέγραψα και αναφέρεται στην βιομηχανική πολιτική που χρειάζεται με τα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας. Επίσης, η τροπολογία 26 έχει το ίδιο πνεύμα. Αναφέρεται στη στήριξη των, ε, στην ανάπτυξη εθνικών επενδυτικών τραπεζών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο ίδιο πνεύμα. Το διαδικό σύστημα σύστημα δηλαδή με θεωρητική μόρφωση και πρακτική εξάσκηση που προτείνει ο κύριος Χατσιμαρκάκης είναι πολύ θετικό. Έχει εμπειρία πολύ καλή η Γερμανία από αυτό το σύστημα και νομίζω ότι θα ήταν καλό να το αξιοποιήσουν και άλλες χώρες. Η κυρία Βάιλερ, την ευχαριστώ ιδιαίτερος για την τροπολογία υπαριθμών ...55... 45 ε, για την ε, πρότασή της και για την κυρία Κόμη και τις τροπολογίες 11 και 45 που ακολουθούν τον ίδιο την ίδια ιδέα ότι δηλαδή δεν μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε άλλες περιοχές του κόσμου, χρειαζόμαστε καινοτομία, χρειαζόμαστε δημιουργικότητα και καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Χέντλ έχει κάνει τροπολογίες που μου φαίνονται ιδιαίτερα ε, συμπαθείς έστω και αν δεν μπορώ με τον τρόπο με τον οποίο τις έχει διατυπώσει να ε, τις υιοθετήσω, να τις συμπεριλάβω στο κείμενο. Θα πρέπει να γίνει κάποια προσαρμογή και για την πιο ισορροπημένη προσέγγιση βιομηχανικής και εμπορικής πολιτικής κλπ. Ευχαριστώ τον κύριο Ροσφόρ, τροπολογίες 6 και 7. Τα μέτρα για την ανάπτυξη και την έρευνα. Και τώρα περνώ στις τροπολογίες στις οποίες έχω κάποιες δυσκολίες. 4, 24, 35, 36, 37 είναι τροπολογίες που πρέπει να Ξανασυζητήσουμε. Πρόκειται για τροπολογίες οι οποίες είτε αποδυναμώνουν το κείμενό μου είτε διαγράφουν κάποια σημαντικά για μένα σημεία. Και πρέπει να πω ότι εδώ έχω προσπαθήσει και για τη βιομηχανική πολιτική να ακολουθήσω μια ολιστική προσέγγιση. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι η πολιτική για τη βιομηχανία δεν είναι απλώς βιομηχανική πολιτική, αλλά και κοινωνική πολιτική και πολιτική καταναλωτού και πολιτική βιωσιμότητας, όπως άλλωστε υπογραμμίζει και με τη τροπολογία της κυρία Πιετικάινεν. Έτσι λοιπόν το να διαγραφούν αυτές οι πτυχές απλά και μόνο ε, δεν βοηθάει γιατί η πολιτική αυτή εξυπηρετεί το συμφέρον του πολίτη, του εργαζόμενου, του εργοδότη, του καταναλωτή. Θέλουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να έχουν σαν αξία ζωής και το περιβάλλον και γι' αυτό δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι αυτοί οι τομείς αποκόπτονται ή αποδυναμώνονται ή και διαγράφονται τελείως από το κείμενο. Εξού και οι τροπολογίες μου με την αρρύθμιση 49 και 40 που στόχο έχουν ακριβώς να ε, ενισχύσουν το κείμενο στο βαθμό που δεν είχα το χώρο στη γνωμοδότηση να συμπεριλάβω. Έτσι λοιπόν έχουμε τον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων, δεδομένων και των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο, πρέπει να πω έχει μεγάλη επικαιρότητα αυτή η πρόταση γιατί εκφράζει πιστεύω ότι, την ιδέα ότι ο πολίτης της Ευρώπης πρέπει επιπλέον να μπει στο, στη γενικότερη κόρα. πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε, όπως είπα, η φορολογική πολιτική και Θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι στο μνημόνιο συνεννόησης και την απόφαση για αύξηση της φορολογίας επιχειρήσεων 10, από το 10 στο 12% έχουμε εντοπίσει σημαντικά προβλήματα προς το συντονισμό και την ισότιμη ή την δίκαιη καλύτερα φορολόγηση ή δίκαιη εξέλιξη ε, τη φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια ιδιαίτερη δυσκολία, την οποία προσπαθώ με την τροπολογία 49 να αντιμετωπίσω. Η δε τροπολογία 40. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε μια περίπτωση που χαρακτηρίζει περισσότερο τη Γερμανία ίσως, Σήμερα στην ε, Γερμανία εορτάζουμε την ε, ημέρα ε, Equal Pay Day, δηλαδή την ημέρα της ίσης αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, γιατί διαπιστώνεται ότι παραμένουν τα προβλήματα και οι ανισότητες στις αμοιβέ μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια πολύ σημαντική πτυχή, μια πτυχή την οποία δεν θέλω να απεμπολίσω και γι' αυτό υπογραμμίζω αυτή την ιδέα της αμοιβή για ισότιμη εργασία. Με την ημέρα αυτή ε, που ερτάζουμε στη Γερμανία και την επικαιρότητά τη, διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκε πρέπει το μήνα να δουλεύουν 8 μέρε περισσότερε, θα έπρεπε μάλλον να δουλεύουν 8 μέρε περισσότερε από ό,τι αντίστοιχα στην αντίστοιχη θέση ένα άντρα για να έχουν τον ίδιο μισθό. Με αυτό το μέλημα καταθέτω τροπολογία υπαριθμών 40 που αναφέρεται στην ε, διεκδίκηση για έναν ελάχιστο νόμιμο μισθό. Ξέρω ότι θα υπάρξουν τροπολογίες, ξέρω ότι θα υπάρξουν αντιπαραθέσεις ε, στο θέμα αυτό και από τους αδέλφους ε, των σκανδιναβικών κρατών γιατί είναι τελείως διαφορετικά τα συστήματα που ισχύουν εκεί. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο του να είμαστε ε, μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μπορεί στα 27 κράτη-μέλη να υπάρχουν είτε ο ελάχιστο νόμιμο μισθό είτε πάρα πολύ ισχυρέ κοινωνικέ ε, συλλογικέ συμβάσει οι οποίε να εξασφαλίζουν το ε, με διαφορετικό τρόπο το ίδιο αποτέλεσμα, το εισόδημα των εργαζομένων και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα θέματα αυτά. Θα προσπαθήσω φυσικά να διατυπώσω συμβαστικέ τροπολογίες με βάση τροπολογίες που κατατίθενται. Ξέρω ότι μπορεί να υπάρξουν ε, διαφορετικές ε, προσεγγίσεις, αλλά θα προσπαθήσω το δυνατόν οι τροπολογίες συμβαστικές να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες. Και πάντως με τι τροπολογίε 1, 2, 8, 9, 10, 31, 32 και άλλες θα προσπαθήσω να διαφυλάξω τη βασική ιδέα της βιομηχανικής πολιτικής από την προοπτική της δικής μας της, κοινοβουλευτική ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ώστε να ενισχύσουμε την έκθεση του κυρίου Λουι Γκρέκ με μια ολιστική προσέγγιση. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέμπχαρτ να μας πούν την άποψή τους οι σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ, λέει η κυρία Κόμη, να ευχαριστήσω την κυρία Κόμη για την, ε, την κυρία Γκέπχαρτ για την εργασία τους. Η βασική θέση της εισηγήτριας βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής και ευχαριστώ τη συνάδελφο ε, για την εργασία της στόχος των δικών μου τροπολογιών και των τροπολογιών του ΕΛΚ αποσκοπούν εις το να αναφέρουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν είχαν σαφώς καταγραφεί και τα οποία κατά την άποψή μας έπρεπε να τύχουν μεγαλύτερης ε, ε, προσοχής εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ με από τα σημεία αυτά. Πρώτα απ' όλα και όπως υπόθηκε έρευνα ε, και καινοτομία θεωρώ ότι για να οικοδομηθεί ε, μια οικονομία βασισμένη στην οικονομική ανάπτυξη, πράγμα που χρειάζεται η Ευρώπη και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη, αυτό είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία ε, που θα πρέπει κυρίως να ενθαρρύνουμε και βεβαίως θα πρέπει να θεωρηθεί και σαν ένα στοιχείο ρόμης για την εσωτερική αγορά. θεωρώ σκόπιμο σημειωθεί και το θέμα της ιχνηλασιμότητας. Ε, είναι σημαντική η ιχνηλασιμότητα για την βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μας δομών, κυρίως αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θυμάμαι τις πρώτες μέρες, ε, τότε που πρωτοεξελέγην ε, βουλευτής και που συζητούσαμε την σήμανση για τα κλωστοϊφανδρουγικά προϊόντα. Εμείς λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ιχνηλασιμότητας ε, για τα προϊόντα αυτά τα οποία πολύ συχνά παραχαράσονται ε, και είναι αποτελέσματα απομίμησης. Ε, κατά αυτήν την έννοια προστατεύεται και ο καταναλωτής αλλά και η βιομηχανία. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω και το οποίο ήδη ευρέως ανέπτυξε η κυρία Γκέπχαρτ είναι ακριβώς αυτό ε, το, είναι το, θέμα της ισότητας των ε, αμοιβών. Ε, η θέση της γυναίκας και εδώ θα πρέπει να διεκδικηθεί και είμαι απολύτως σύμφωνη. Επίσης, η πραγματική μισθή. Δεν θέλω τώρα να μπω ε, στο θέμα της ε, δυναμικής ε, της ελευθερίας που μπορεί να έχει κάποια επιχείρηση όσον αφορά τις αμοιβέ των εργαζομένων. Επομένως, άλλο είναι η ισότητα των φύλων και άλλο αυτό το ζήτημα. Το να επιβληθεί ε, μία ή μία ε, εξίσωση των ε, μισθών πιστεύω ότι δεν είναι ο σωστός δρόμος γιατί θα πρέπει αυτοί οι μισθοί να αποτελέσουν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορέσουμε κατά την άποψή μου να ξανασυζητήσουμε δελεχέστερα. κάτι άλλο το οποίο με αφήνει λίγο με ερωτηματικά ε, είναι, αυτά το, είναι το θέμα των βιομηχανικών πάρκων. Εγώ συμφωνώ με τα κλάστερς και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο διαμονής συγγνώμη, διανομής βελτιώνουν τις συνέργειες, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην σύνθεση ε, που ε, θα έχουν τα κλάστερ, γιατί ε, ενδεχομένως θα δημιουργηθούν κάποιες συνέργειες αρνητικές, οι οποίες θα δημιουργήσουν τελικά πρόβλημα στην εδαφική επικράτεια στην οποία να βρίσκονται. Θα πρέπει λοιπόν τα κλάστερ να βρίσκονται σε στενή επαφή με την περιφέρεια. Εγώ ας πούμε σκέφτομαι τα κλάστερς τα οποία έχουν δημιουργηθεί ε, και για την κλωστοϊφαντουργία και για τις ε, νέες ε, τεχνολογίες. Εκεί δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή προσωπικού. Επομένως, ναι, βεβαίως να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, αλλά θα πρέπει ε, να προστατέψουμε και αυτούς ε, που θέλουν να εξακολουθήσουν να δουλεύουν στην περιοχή τους ή στην εταιρεία, στην επιχείρηση στην οποία ξεκίνησαν πριν από χρόνια να δουλεύουν. Είμαι επεπισμένη πάντως ότι η συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα και ε, η επικοδομητική ανταλλαγή ε, των απόψεών μας ε, ταυτίζεται με την γενική αρχή ε, που λέει ότι για να υπάρξει ανάπτυξη της βιομηχανίας θα πρέπει να υπάρξει και ανάπτυξη της της επιχειρηματικότητας. Ε, όσον αφορά τώρα τις ε, καθυστερημένες ε, καταβολές χρημάτων αμοιβών από το δημόσιο. Στη χώρα μου αυτό ισχύει και εάν τα χρήματα είχαν ε, δοθεί στην ώρα τους θα είχαν ε, δημιουργηθεί γύρω στις 250.000 ε, θέσεις εργασίας. τι να σας πω τώρα, στην Ευρώπη έχουμε μάθει να μην δουλεύουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Εδώ όμως αυτό δεν συνέβη. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη η έγκριση και η υιοθέτηση της οδηγίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ε, και η μεταφορά στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών. Και βεβαίως μετά η θέση σε ισχύ, η επικύρωση των κρατών μελών ε, είναι πολύ σημαντικά θέματα. Και μια τελευταία σκέψη. Στη χώρα μου δεν υπάρχει κυβέρνηση και βρισκόμαστε σε μια ε, στάσιμη ε, περίοδο και αυτό βαραίνει ιδιαίτερα την βιομηχανία και τη βιομηχανική πολιτική. Επομένως τέτοιες πολιτικές μπορούν να ξεκουνήσουν λίγο την κατάσταση και να κάνουν καλό και στη χώρα μου αλλά και στην, Ιταλία, στην Ευρώπη στο ευχαριστώ. κύριος Χατζημαρκάκης, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, σε αυτά που και η κυρία Κόμη θα συμφωνήσω και στα όσα είπε η κυρία Γκέμπχαρτ ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια πιο ισότιμη κατανομή της εκβιομηχάνησης στην Ευρώπη. Χαίρομαι που δέχεται τις τροπολογίες μου η κυρία Γκέμπχαρτ. Εδώ βρισκόμαστε και στο επίκεντρο της συζήτησης, της επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ε, επιβάλλουμε στον Ευρωπαίο κατά τρόπο νέο υπεριαλιστικό θα έλεγα τι είναι καλό και τι είναι σωστό και τι πρέπει να κάνει και ταυτόχρονα να μην του επιτρέπουμε μια ισότιμη ανάπτυξη της βιομηχανικής πολιτικής και να αποκλείονται από, τη το βιομηχανικό σχεδιασμό ολόκληρες περιοχές της Ευρωζώνης. Αυτό λοιπόν νομίζω δείχνει ότι είναι σωστή η κατεύθυνση την οποία ακολουθεί η κυρία Γκέπχαρτ και τη συγχαίρω ο σχετικά περιορισμένος αριθμός των τροπολογιών μας δείχνει άλλωστε ότι ήταν ε, από την αρχή ε, καλά σταθμισμένο το κείμενο, διαφορετικά θα είχαν κατατεθεί πολύ περισσότερες τροπολογίες. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ωστόσο για την τροπολογία 43, τη διαδική εκπαίδευση-κατάρτιση, δηλαδή εκπαίδευση και ε, επαγγελματική εκπαίδευση ή εξάσκηση, ε, ότι χρειάζεται για τους νέους να έχουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση. Ε, η Ισπανία μπορεί να έχει μια καλή, κάποιες καλές επιδόσεις, αλλά η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα έχει τραγικά στοιχεία ως προς την επαγγελματική κατάρτιση των νέων, την εκμάθηση ουσιαστικά. Και νομίζω ότι σε αυτό θα μπορούσαμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα της Γερμανίας ε, και γι' αυτό καταθέτω την τροπολογία 43, που θεωρώ ότι πρέπει να συνδυαστεί στενά με την βιομηχανική πολιτική, γιατί δεν μπορεί δεν αρκεί να έχουμε μόνο βιομηχανική πολιτική, αλλά ποιοτική κατάρτιση, επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί αυτό ουσιαστικά επιδιώκει, αυτό ουσιαστικά επιτυγχάνει το διαδικό σύστημα στην εκπαίδευση. Πιστεύω ότι θα βρει πλειοψηφία και ελπίζω ότι θα την υποστηρίξουν όλοι οι συνάδελφοι την κυρία Γκέπχαρτ. Ε, πάντως ήταν πολύ καλό το κείμενο. Ευχαριστώ. Κυρία Ρούλε δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλος το λόγο. να πω και εγώ δύο λόγια, θα συμμετάσχω και εγώ στη συζήτηση. Συμφωνώ με την γενική πορεία της συζήτησης. Αναφέρθηκε η σημασία μιας βιομηχανικής, μιας ολιστικής ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής και εν ώψη του ορίζοντα 2020, αλλά και στα θέματα των δημοσίων προμηθειών που καλύπτουν κάποιες τροπολογίες. Ε, κυρία Γκέπχαρτ, ε, υπάρχουν πρόσωποι της Επιτροπής εδώ, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Με ένα λεπτό. Η κυρία Λουγκρίπ θέλει το λόγο. Με συγχωρείτε, δεν σας είχα δει στον κατάλογο, παρακαλώ. Εγώ αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό είναι που συζητάμε για τη βιομηχανική πολιτική για την Ευρώπη, είπε η συγγετρία κυρία Γκέμπχαρτ, έτσι μας είπε και χαίρομαι πάρα πολύ καλά που το είπε. Ε, βιομηχανική πολιτική λοιπόν ε, είπε και χαίρομαι που δεν είναι πια λέξη ταμπού όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια. Τουλάχιστον εδώ στις βρυξελιώτικες ε, περιοχές. επιμένει η συγκήτρια ανάμεσα στην ανάκαμψη της βιομηχανίας στην Ευρώπη ε, και την εφαρμογή, την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς. Εγώ συμμερίζομαι πολύ τον, πολιτι... τον προσανατολισμό αυτό και αυτή την προσέγγιση. Για να μπορέσουν ε, οι ευρωπαϊκές βιομηχανικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν, και για να βοηθήσω στη διαδικασία υπέβαλα κάποιες ε, τροπολογίες τις οποίες κάποιοι συνάδελφοι ε, είχαν την καλοσύνη να προσυπογράψουν ε, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης νησίας αγοράς μιας γρήγορης και αποτελεσματικής εφαρμογής της εφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας την υλοποίηση της Small Business Act που αφορούν την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που ε, πρέπει να είναι σαφώς συνδεδεμένη με μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική, βεβαίως ενισχυμένη συνεργασία ε, ε, από την αρχή της διαδικασίας με εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων, που αυτό είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για μεταφορά και υλοποίηση των ενωσιακών νομοθεσιών, νομοθετημάτων μάλλον. Νομίζω ότι με σωστό και διορθωμένο τρόπο πρέπει να στείλουμε ένα καλό μήνυμα σε έναν ικανό και με καλή επίδοση ε, ευρωπαϊκό τομέα που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ε, ε, σαν τομέα αριστείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν μέσω μιας τροπολογίας να υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να βοηθηθούν αυτές οι βιομηχανίες της ευρωπαϊκής αριστείας που τα μάλα συμβάλλουν στην ανάπτυξη στην ε, ε, ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3% του ΑΕΠ με 100 δις ευρώ κύκλο εργασιών έχουν αυτές ε, οι επιχειρήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως έχουν σημαντικό οικονομικό και εμπορικό βάρος. Από την άλλη πλευρά πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες ε, είναι στραμμένες προς την εξαγωγή, οι οποίες αναπτύσσονται, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στις πολύ σημαντικές επιχειρήσεις, τα μεγάλα ονόματα, τα βαριά, τα οποία όλοι φέρνουμε στο νου μας όταν αναφερόμαστε σε Οντεγκάμ και σε ε, ε, ε, Αριστεία. Αναφέρομαι σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες ε, ασχολούνται με την διατήρηση των παραδόσεων, τη διατήρηση των παραδοσιακών γνώσεων, ε, αυτές οι οποίες άμεσα συνδέονται και αποτελούν το ενωσιακό ευρωπαϊκό ε, ε, παρελθόν, την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Ancré dans l'histoire européenne depuis euh, de, nombreux siècles, euh, un art de vie. Και νομίζω ότι είναι αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες μεταφέρουν ένα σύστημα αξιών, ε, μία συγκεκριμένη ιδέα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να ζούμε, του, του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αναπτυσσόμαστε, του τρόπου με τον οποίο πρέπει να διατηρούμε τις παραδόσεις μας. Ε, και βεβαίως πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να ε, μεταθέσουν γεωγραφικά τις ε, δραστηριότητές τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι αυτοί οι τομείς του αυτό, αυτοί οι τομείς λοιπόν της Ευρωπαϊκής Αριστείας είναι οι τομείς οι οποίοι δημιουργούν θέσεις εργασίας, οι οποίοι έχουν εργαζόμενους ικανοποιημένους, είναι αυτοί οι οποίοι απασχολούν τεχνίτες, τεχνίτες με παραδοσιακές γνώσεις, ε, που ε, μεταλαμπαδεύουν στους νεότερους ε, συγκεκριμένες γνώσεις οι οποίες είναι παραδοσιακές και που δεν πρέπει να χαθούν, επαγγέλματα που δεν πρέπει να χαθούν. Από το Σεπτέμβριο του 2012 είχαμε μια ανακοίνωση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την, ε, για την υψηλού επίπεδου ευρωπαϊκή βιομηχανία, την βιομηχανία Odegam και αριστείας και στην ανακοίνωση αυτή ανεγνώριζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη σημασία και το βάρος του κλάδου αυτού. Και επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά ότι στον κλάδο αυτό έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά έχουμε και ένα μεγάλο δίκτυο μικρομεσαίων μεσαίων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια που ε, πρέπει να αντιμετωπιστούν βάσει των εξειδικευμένων τους αναγκών και βεβαίως ε, με εξειδικευμένο τρόπο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους τα οποία σχετίζονται με την παραχάραξη, με την απομίμηση. Ε, όλα αυτά θα πρέπει να τα ξαναπούμε και θα πρέπει να δώσουμε όλη μας την προσοχή σε αυτόν τον τομέα ο οποίος για μία ακόμα φορά λέω ότι είναι στραμμένος προς τις εξαγωγές και ότι είναι ένας εξαιρετικά υγιής κλάδος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε χρόνο. Έχετε παρακολουθήσει το θέμα από κοντά, οπότε έχετε ένα λεπτάκι αν θέλετε να υποβάλει κάποια παρατήρηση. Uh, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές στην Επιτροπή, διότι ε, αποδοστολθεί τη σημασία στην ανακοίνωσή μας. Μιλούμε τώρα για την βιομηχανική πολιτική. Όχι μόνο ασκούμε τέτοια πολιτική, αλλά αυτά όλα τα επιμέρους στοιχεία τα οποία περιέχονται στην ανακοίνωση τώρα τα επεξεργαζόμαστε και υπάρχει και για τις υπηρεσίες ε, των επιχειρήσεων έχουμε μία ομάδα υψηλού επίπεδου, έχει συγκροτηθεί, αποδίδει για τις επιχειρήσεις και θεωρούμε ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας για τον κλάδο των υπηρεσιών, τον κατασκευαστικό και θέλουμε έτσι οι επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν εισρωή ρευστού. Να μπορούν να αυτοχρηματοδοτούνται. Και πολλές φορές αυτή η εισρωή χρημάτων ε, πολλές φορές όπως και στη δική μου χώρα σταματά ακόμα για 800 μέρες. Επομένως το θέμα δεν είναι απλώς οικονομικό. Είναι και κοινωνικό. Οπότε πρόκειται και για κοινωνική πολιτική που θα πρέπει εν προκειμένου να χαράξουμε. Κάτι να προσέξετε στην τροπολογία βαθμών 5, εκεί γίνεται η μνήμα της επιλογή των 6 αγορών. Όχι, αυτό είναι λάθος. Είπαμε για έξι τομεί που θα τύχουν υψίστες προτεραιότητε. Αυτά θέλουμε να απασχολήσουν την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση και για νομοθεσία, πρότυπα και για ε, διάφορα μέτρα και μέτρα εξωτερικής πολιτικής, διότι πρόκειται για κάποιες αγορές που είναι νέες, αναπτύσσονται και θα μεγαλώσουν ταχαίως τα μέσα επόμενα χρόνια. Επομένως δεν είναι έξι, έξι αγορές, είναι έξι τομείς. Ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω τώρα θέλει η συγγήτρια να ολοκληρώσει. Νομίζω 24 Απριλίου θα ψηφίσουμε. κυρία Γκέπχαρτ, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Ναι, σύντομα. Δύο-τρεις παρατηρήσεις. Καταρχάς, πρέπει να προσέξουμε να μην κάνουμε πολύ μεγάλη εξειδίκευση στη βιομηχανική πολιτική, δηλαδή να μην αποτρέψουμε, να μην κλείσουμε το δρόμο σε νέες εξελίξεις που ενδεχομένως δεν έχουμε κάνει υπόψη μας ακόμη. Δεν μπορούμε δηλαδή να περιγράψουμε αυστηρά και άτεγκτα τους τομείς έτσι ώστε τελικά να κλείσουμε ευκαιρίες που ενδεχομένως να υπάρχουν. Πρέπει να αφήσουμε ένα περιθώριο ευελιξίας και να δούμε τι είδους νεοτερισμοί υπάρχουν, τι είδους καινοτομίες, δημιουργικότητα μπορεί να αναπτυχθεί. Και γι' αυτό, για την κυρία Λουκρύπ και την κυρία Κόμη, δεν θέλησα να καταγράψω κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Εσείς μιλάτε για το αρτιζανά, τη βιοτεχνία, η κυρία Κόμη βεβαίως για τη ε, φαντουργικά. Εγώ θα μιλούσα ίσως για αυτοκίνητα και ε, βαρύ εξοπλισμό, ε, βαρέα βιομηχανία. Ναι, αλλά έτσι εξειδικεύουμε υποχρεωτικά και αποκλείουμε υποχρεωτικά κάποιους τομείς. Γι' αυτό θέλω να αποτρέψω αυτού, αυτές τις διευκρινήσεις. Γι' αυτό θέλω η βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη και στην περιφέρεια, όπως επεσήμανε πολύ σωστά ο κύριος Χατζημαρκάκης, να έχει την ευκαιρία στην ανάπτυξη χωρίς αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ βιομηχανικών ζωνών και χωρίς να ε, δούμε μετατόπιση βιομηχανικών δραστηριοτήτων από τη μία περιοχή στην άλλη, γιατί είναι πιο ευνοϊκή η όρη. Αυτό θέλω να καταστήσω απόλυτο σαφέ. Για τον κύριο Χατζημαρκάκη δεν χρειάζεται. Κύριε Χατζημαρκάκη, εμένα να με πείστε για το διαδικό σύστημα. Ε, θεωρώ ότι είναι πάρα, πάρα πολύ καλό. Εγώ έχω μεγαλώσει στη Γαλλία και βλέπω τι διαφορέ μεταξύ των δύο συστημάτων. Το διαδικό σύστημα τη Γερμανία με την ε, ε, ε μαθητεία, την, την επαγγελματική ε, κατάρτιση δίνει και στην πρακτική τη δυνατότητα στον νέο να υλοποιήσει αυτά που θεωρητικά έχει μάθει. Είναι πάρα πολύ καλό λοιπόν και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και αν δεν με ακολουθήσει λοιπόν η ομάδα μου, αν και είμαι βεβαίω ότι θα με ακολουθήσει, η, την τροπολογία σας, την 43, θα την συμπεριλάβω στο κείμενο οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα γίνει λοιπόν η ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση και τις συμβαστικές αστροπολογίες στις 24 Απριλίου και συνεχίζουμε με μια συζήτηση για ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα για την οδηγία προ... τη σχετική με τα προϊόντα καπνού. Κυρία Χάντσλικ. Θα, θα, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Χάντσλικ να μας κάνει την παρουσίαση και αναλόγως θα προσανατολιστούμε για ένα πρώτο χείρο συζητήσεων. Επαναλαμβάνω βεβαίως ότι μας πιέζει ο χρόνος. Κυρία Χάνσλικ. Και νομίζω έχουμε τον κύριο Σεσέλ εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναπληρωτής ε, διευθυντής της ΑΝΚΟ. Ο κύριος Ρή είναι ο διευθυντή. Με συγχωρείτε, λάθο σημείο διάβαζα. Αν πάση περιπτώσει, σας καλωσορίζουμε. Θα ακούσουμε την παρουσίαση σε λίγο, αλλά πρώτα την κυρία Χάνσλικ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Στόχος της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού είναι να βελτιωθεί η εσωτερική αγορά ε, μέσα με ταυτόχρονα όμως προστασία των καταναλωτών και της υγείας τους. Η Κομισιόν λέει ότι δεν θέλει να επικεντρωθεί μονάχα ε, στους ε, παρόντες καπνιστές. Λέει ότι θέλει να μειώσει την ελκυστικότητα των προϊόντων καπνού έτσι ώστε οι νέοι και κυρίως οι νέοι χρήστες και κυρίως οι νέοι στην ηλικία χρήστες να μην θέλουν πλέον να έχουν το πακέτο των τσιγάρων δίπλα Πρόκειται για μια στάση την οποία να συμμερίζομαι απολύτως. Η Κομισιόν ε, υποβάλλει διάφορες ε, καλές ε, λύσεις αλλά και κάποιες άλλες οι οποίες με αμφίνουν λίγο με, σε αμφιθυμία. Ε, ακριβώς αυτά θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε, αυτά τα σημεία, γιατί σύντομα θα μας παρουσιάσει η Κομισιόν ε, και μία μελέτη αντικτύπου, ε, η οποία φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μεγάλη επικέντρωση προσοχής δείχνει η Κομισιόν στην συσκευασία γιατί πρέπει να είναι αποτρεπτική η συσκευασία ε, και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να οδηγηθεί κάποιος και στο κόψιμο του, του καπνίσματος ε, λόγω της αλλαγής της συσκευασίας. Ας πούμε... Ε, υπάρχουν κάποιες συσκευασίες που θυμίζουν κατά κάποιο τρόπο, τι να σας πω, ένα κραγιόν ας πούμε. Αυτές πρέπει οι συσκευασίες να απαγορευτούν. Ε, βάσει των ε, στοιχείων του Ογκολογικού Κέντρου της ε, Βαρσοβίας περί τα τέλη της δεκαετίας του 90 που είχαν σκοπό να μελετήσουν τον αντίκτυπο των τεστ, μάλλον όχι των κειμένων και των λεκτικών προειδοποιήσεων στην Πολωνία, σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, ε, λέω, 4% ε, των ε, καπνιστών στη χώρα μου σταμάτησαν να καπνίζουν λόγω ακριβώς αυτών των κειμένων, των προειδοποιητικών και αποτρεπτικών του καπνίσματος και ένας άλλος αριθμός καπνιστών προσπάθησε να κόψει το τσιγάρο έστω και αν τελικά δεν το κατάφερε. Είναι πολλοί οι Πολωνοί, οι οποίοι η πλειοψηφία των Πολωνών ε, είπαν ότι μπορούν πραγματικά αυτά τα προειδοποιητικά κείμενα να είναι αποτρεπτικά ε, για το κάπνισμα. Θα πρέπει βεβαίως να έχουμε την δυνατότητα να δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν αυτά τα αποτρεπτικά κείμενα στο άρθρο 6 γίνεται λόγος και για τον ε, όγκο που θα πρέπει ή την επιφάνεια που θα πρέπει να καλύπτουν ε, αυτά τα προειδοποιητικά κείμενα. Επίσης ε, γίνεται λόγος για τις αρωματικές ουσίες, δηλαδή εάν είναι ένα επιπλέον εθιστικό στοιχείο η συμπερίληψη τέτοιων αρωματικών ουσιών. λέμε ότι οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες στην Ευρώπη και να έχουν παρόμοια προειδοποιητικά στοιχεία. Αυτό είναι κάτι καλό. όλοι συμφωνούμε ότι το τσιγάρο καλό πράγμα δεν είναι. Όμως τι, σε τι μπορεί να ε, συμβάλλει η απαγόρευση συμπερίληψης αρωματικών ουσιών εάν τα τσιγάρα μπορούν να, ε, ε, να πουλιούνται. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτή η ιδέα για τις αρωματικές ουσίες να έχουν ένα συγκεκριμένο αντίκτυπο. Λοιπόν, εδώ θα θέλω να σας ε, δείξω ένα πακέτο ε, παράνομων τσιγάρων. Εάν, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, απαγορεύσουμε τελείως αρματικές ουσίες, μπορεί να συμβεί το εξής. Αυτή τη στιγμή μπορεί κανείς να αγοράσει ένα παράνομο πακέτο τσιγάρων. Εγώ έχω ένα τέτοιο παράνομο τσιγάρο, σας το δείχνω τώρα. Και ε, ακριβώς χάρη σε τούτο το πακέτο μπορεί κανείς να ε, ε, κατασκευάσει ένα τσιγάρο με, με, με, με μαντόλ. Δηλαδή, απλώς παίρνετε το τσιγάρο, και παίρνετε και αυτό το σπρέι με το μεντόλ και ε, ε, πρέπει να σας πω ότι βρωμάει φρικτά, δεν έχει καμία σημασία, εγώ θεωρώ ότι βρωμάει. Είναι μία αηδία, επιτρέψτε μου να σας πω. Πάντως, πραγματικά, ε, αυτά τα τσιγάρα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, για όλη τη βδομάδα, θα κρατήσουν αυτήν, αυτό το άρωμα της, του, του μεντόλ. Και επομένως, εάν από τη μία μεριά απαγορεύσουμε τσιγάρα με μεντόλ, Απ' την άλλη πλευρά όμως εξακολουθούμε να επιτρέπουμε την πώληση των σπρέι μεντόλ, τότε δεν έχουμε, δεν καταφέρνουμε να κάνουμε κάτι. Ναι, ναι, βρωμάει, το ξέρω κύριε Πρόεδρε και εσείς τώρα το μυρίζετε και βλέπετε. Κοιτάξτε, ε, ε, αυτό το άρωμα κυρίες και κύριοι έχω κάνει το πείραμα στο σπίτι μου, θα κρατήσει για δύο εβδομάδες τουλάχιστον. Επομένως, τι να κάνουμε, έχει έννοια να ε, αποκλείσουμε και τα αρώματα, αυτές τις αρωματικές ουσίες στην αγορά. Όχι, δεν έχει έννοια. Επομένως, τι να σας πω. Επίσης, ε, ε Έχουμε και άλλο προβληματισμό όσον αφορά ας πούμε την ε, ε, εξαποστάσεως ε, πώληση μέσω ίντερνετ κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παραστατικά μας το είπατε. Να, ναι, εδώ είναι, εδώ είναι το καταγραφεί και από την κάμερα. Αυτά, super slim. Αυτά υποτίθεται έχουν επαγορευτεί. Από πού τα αγοράσατε, από πού προέρχονται. Στο Μίνσκ, ε. Καλά. Okay. Um... All right. Well, look, um, uh, I'm... Πρόεδρος. Δώρο, δωράκι του Λουκασέγκο. Let's, um, ask, let us ask the commission. Για να απευθύνουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας ε, παρουσιάσει τι έχει σε σχέση με αυτό το σημαντικό ζήτημα, κύριε Ρίς. Ποια είναι η στρατηγική σας σε σχέση με την αναθεώρηση του νομοθετήματος. Very much, ε, Η Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε αυτή την παρουσίαση την 20η, οπότε ε, να εξασφαλίσουμε και λίγο χρόνο που να σε η συζήτηση. Έχουμε εδώ πέρα διάφορα ενδιαφέροντα προϊόντα που θα μπορούσα να σας ε, παρουσιάσω αλλά όλα αυτά θα τα στήσουμε μπροστά στις κάμερες στο τέλος παρουσίασης. Όταν ξεκινήσαμε την διαδρομή αυτή, η οδηγία εγκρίθηκε το 2001. Από τότε έχουμε μια σειρά εξελίξεων, νέα προϊόντα, νέα στρατηγικές. Όπως και η εισηγήτρια είπε ε, new scientific Έχουμε επομένω τώρα στοιχεία επιστημονικά. Δεκαετία του 70 ξεκίνησε η έρευνα και στη ΣΥΠΑ είχαμε την πρώτη έρευνα σε σχέση με το ότι το κάπνισμα σκοτώνει για τον καρκίνο και τότε άρχισαν οι επιστημονικές επιτροπές να μελετούν και τις επιπτώσεις στην υγεία αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Έχουμε γνωστρά όλες αυτές τις μελέτες σε πολλές χώρες και έτσι μπορούμε να τα λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία ως Ευρωπαϊκή Ένωση λάβαμε κάποιες πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις όταν αποφάσαμε να προσχωρήσουμε ε, στο, στα μέτρα που ο ΠΟΕ έλαβε για τον έλεγχο των προϊόντων καπνού και, τα, κάποια μέλη τέλο πάντων ρέψαν ε, έντονη δραστηριότητα. Γιατί φυσικά με το προσχώρησε κανείς αυτή την συνθήκη ανέλαβε και κάποιες υποχρεώσεις. Και ε, τώρα, η αγορά και το προϊόντα το καπνό. Πώς είναι το τοπίο σήμερα. Δεν ξέρω αν μπορεί να διακρίνεται τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά τέλος πάντων θα διαβάσουμε στη γραμματεία τα σχετικά έργα που θα πάρει από εκεί. Το κυρίαρχο προϊόν στην αγορά είναι τα τσιγάρα. 89% της αγοράς και ο καπνός για στρίψιμο είναι το 7% της αγοράς. η αξία σε χρήμα βλέπουμε τα στοιχεία του 2010. Είναι βέβαια και τα έσοδα από την φορολόγηση. και βλέπετε τα στοιχεία όσον αφορά τα, τα, τα, τα χρήματα, όσον αφορά τα οικονομικά και για τον καπνό, για στρίψιμο. 42% είναι η μεταβολή. Καπνός τώρα για πίπα. Εκεί έχουμε μείωση. Ε, difficult to explain because was a change in the, in the... Βλέπουμε εδώ πέρα τη μεταβολή όσον αφορά τις πωλήσει. Έχουμε και στην ονοματολογία κάποιες αλλαγές ε, που, που, έχουν γίνει. Βλέπετε και για τα σιγαρίλος και για τα πουρα. Εδώ η αγορά είναι μικρότερη και μετά πάμε στην ε, ανάλυση των κινδύνων για την υγεία και τις οικονομικές επιπτώσεις. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα γίνουν λιγότερο ελκυστικά αυτά τα προϊόντα για τους νέους. Πότε αρχίζει κανεί το κάπνισμα. Στην Ευρώπη πολλοί αρχίζουν να καπνίζουν αρκετά νέοι. στα 15, στα 18, 70% των καπνιστών αρχίζουν πριν φτάσουν τα 25, 95% και 70% πριν τα 18. Επομένως αυτή, αυτή είναι η ομάδα ε, που στοχεύουμε με αυτά όλα τα μέτρα. Αλλά βέβαια σε αυτού στοχεύει και η καπνοβιομηχανία. Και είναι για την υγεία. Έχουμε περίπου 70. 700.000 περίπου όσοι κατοικούν στη Φραγκφούρτη πεθαίνουν από την χρήση τέτοιων προϊόντων καπνού. Αν δεν κάπνιζαν, μπορεί να σωζόντουσαν. Οι επιδημιολόγοι έτσι κάνουν τον υπολογισμό και επομένω υπολογίζουν οι επιδημιολόγοι ότι αυτό αντιστοιχεί σε 8,5 εκατομμύρια έτη ζωής. Θα μπορούσαν, υπολογίζεται, να ζούσαν ακόμη 14 χρόνια οι καπνιστές. Και η δαπάνη όσον αφορά τις ιατρικές αγωγές για τις βλάβες από το κάπνισμα η δαπάνη ανέρχεται στα 25,3 δις ευρώ. Η δε κοινωνία χάνει ετησίως 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ από πλευράς ε, απώλειας παραγωγικότητας. Άρα θα πρέπει να έχουμε περισσότερα χρόνια με υγεία, περισσότερο εργατικό δυναμικό, το να είναι υγεία. Έχουμε τώρα τι μέτρα προτείνουμε. Πρώτα απ' για τα περιεχόμενο. Θέλουμε να αναβαθμιστούν οι υποχρεώσεις κοινοποίησης σε σχέση με την ε, τρέχουσα, ισχύουσα οδηγία δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Απαγόρευση για τα τσιγάρα. Τα τσιγάρα, τον καπνό για στρίψιμο με κάποιες ε, γεύσεις και αρώματα. Γιατί εδώ υπάρχει υυξημένος κίνδυνος εξάρτησης και τοξικότητας. Αυτά τα πρόσθετα τα οποία μερικά συνεχίζουν να επιτρέπονται όσον αφορά τη χρήση τους. Συσκευασία και ετικετοθεσία. Υποχρεωτική προειδοποίηση με μια μεγάλη ε, φωτογραφία, γραφική παράσταση και στις δύο πλευρές. Εάν τελικά εγκριθεί η πρόταση, και να καλύπτει 75% του πακέτου και στις δύο πλευρές. Του πακέτο αλλά και της συσκευασία του καπνού για στρίψιμο. Απαγόρευση των τσιγάρων slim. μπορούν τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν συσκευασία χωρίς παραστάσεις. Εάν είναι αυτό, συμβατό προς την συνθήκη και αιτιολογείται ειδικά. Η ισχύουσα οδηγία επιτρέπει τις επισημάνσεις, τις προειδοποίησεις με γραφική παράσταση, με εικόνα αν έχει οψιμότητα έχει λασιμότητα, θα πρέπει αυτό να ισχύει μέχρι τον πρώτο λιανοπολιτή. Και θα πρέπει σε όλες τις συσκευασίες να πάρουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας Ούτω ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσον υπάρχει κάποιο είδου απομίμηση ε, γιατί το προϊόν είναι γνήσιο. Επίσης, θέλουμε να συνεχίσει η απαγόρευση του καπνού που ε, ρουφάμε από τη μύτη. Αυτό αφορά την Σουηδία κυρίως. Επίσης ε, και στις δύο πλευρές της συσκευασία και να μην έχουμε αυτές τις ε, ιδιαίτερες ε, γεύσεις για αυτά τα προϊόντα. Όσον αφορά τις πωλήσει από απόσταση, τις διασυνοριακές, εδώ χρειάζεται κοινοποίηση και έγινε και μελέτη επιπτώσεων ε, όσον αφορά τις πωλήσει από το διαδίκτυο και γι' αυτό αποφασίζαμε να λάβουμε αυτό το μέτρο. Τώρα όσον αφορά τα καινούργια προϊόντα, τα οποία τώρα αναπτύσσονται, εξελίσσονται, θέλουμε αυτά να κοινοποιούνται και αυτό να είναι υποχρεωτικό. Και συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις της ισχυρής οδηγίας TPD. Τώρα, για τα ηλεκτρικά τσιγάρα και συναφή προϊόντα, ηλεκτρονικά τέλος πάντων, εδώ θέλουμε να ισχύσει το κατόφλι, επί του καθορίζεται το κατά πόσον αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τη σχετική νομοθεσία που ήδη ισχύει. Αυτό ισχύει και για τις ε, ε, τσίχλες, ε, για αυτά τα, τα, αυτοκόλλητα, τα πάτσες. σε σχέση και με την νομοθεσία για φαρμακευτικά προϊόντα. Επίσης, θεσπίζονται κανόνες για την κατοθεσία και προειδοποιήσεις όσον αφορά τα φυτικά προϊόντα που καπνίζονται. Να βλέπετε τώρα πώς θα είναι το πακέτο με αυτές τις ε, παραστάσεις, πώς θα είναι στο μέλλον. Όσο αφορά τώρα, τελικά, με τις δύο τελευταίες διαφάνειες όσον αφορά τις επιπτώσεις της κοινωνικο-οικονομικές της αναθεώρησης του νομοθετήματος, ε, ε, ρίξω μια ματιά όσον αφορά τον συνδυασμό των προτιμωμένων επιλογών πολιτικής. Θέλουμε σε πέντε χρόνια να έχουμε ε, μείωση στην κατανάλωση προϊόντων καπνού κατά 2%. Δεν είναι τόσο φιλόδοξο στόχος αυτός, μερικοί μας λένε, αλλά θεωρούμε ότι είναι αξιόλογος στόχος. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα έχουμε μείωση των καπνιστών κατά 2,4 εκατομμύρια. Ε, οι πιθανές ζημίες για την καπνοβιομηχανία θα αντισταθμιστούν από τα μέτρα που θα λάβουμε κατά του λαθρεμπορίου ή του παρανόμου μπορεί το πάντων. Και βέβαια τα χρήματα τα οποία τώρα κανείς ξοδεύει σε προϊόντα καπνού θα μπορεί να τα ξοδεύει σε κάτι άλλο. Τα ωφέλη. Θα ζει κανείς περισσότερα χρόνια, θα έχει καλύτερη υγεία, μιλάμε για 9,4 ε, δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως ως εξοικονόμηση, ε, μείωση των δαπανών υγείας κατά 506 εκατομμύρια και μείωση των ε, απολειών από την λιγότερη παραγωγικότητα κατά 165 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε επομένω αυτό το 2% που να μειώσουμε και οπότε θα έχουμε 1,59 δις ευρώ όσον αφορά του λιγότερους φόρους και ε, αυτό θα αντισταθμιστεί από μια αύξηση των φορολογικών συντελεστών σε αντίστοιχους φόρους που επιβάλλονται. Μπορείτε εδώ πέρα αυτό να στον ιστότοπο και επίσης μπορούμε να σας ε, ε, απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις όπως είπε και η, ε, Και έχουμε και εκατοντάδες επιστημονικών άρθρων όσον αφορά τις επιπτώσεις του καπνίσματος. Τώρα θα σας δείξω ορισμένα προϊόντα για να καταλάβετε τι μεταβολές θα γίνουν. Πάμε στις επόμενες διαφάνειες. Oh, Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε χρόνο δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Τι, πώς να σας το πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βλέπω κάτι χέρια που σηκώνονται εδώ. Έχω κάποιου γραμμένους στον κατάλογό μου, Επομένω θα πρέπει να του δώσω το λόγο. Γκέμπχαρτ Μάγερ, παρακαλώ πολύ, μην πολύ μιλήσετε, γιατί πρέπει να τελειώσουμε στην ώρα μας. Ε, καλό θα ήταν ίσως να ασχοληθείτε και με κάποια από τα σημεία της ε, εισηγητρίας. Στάιλερ Σμιτ, Μπίτ, να μην ε, μιλήσετε πάρα πολύ ώρα ο καθένας, μερικά λεπτά μόνο. Θα έχουμε αργότερα τη δυνατότητα να κάνουμε και ε, πιο αναλυτικές ε, παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ και την Κομισιόνα για την εντελεχή παρουσίαση. Είμαι και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και δουλεύουμε για την αναθεώρηση της οδηγίας βάσει της οποίας θα υπάρχουν και εικόνες ε, στις συσκευασίες των τσιγάρων. Νομίζω ότι η αλλαγή της συσκευασίας είναι πάρα πολύ καλή. 30 εκατομμύρια ε, άνθρωποι υποφέρουν ε, κάθε χρόνο από τις επιπλοκές ε, της υγείας τους λόγω της κατανάλωσης προϊόντων καπνού και πάρα πολλοί είναι αυτοί που χάνουν και τη ζωή τους. Καλωσορίζω λοιπόν τις προτάσεις της ε, Κομισιόν. Νομίζω ότι η αναθεώρηση είναι μια καλή ευκαιρία. Στηρίζω λοιπόν ε, τις ε, προτάσεις βάσει των οποίων 75% της επιφανίας της συσκευασίας θα πρέπει να καλύπτεται από προειδοποιήσεις υγείας αλλά θέλω να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Ε, βεβαίως ε, η προσθέμενη αξία είναι για τις βιομηχανίες καπνού η φύρμα. Εάν αφαιρέσεις τη φύρμα τότε αφαιρείς και αυτήν την κορυφή του παγόβουνου που είναι ορατή. Επομένως η συσκευασία πρέπει να παίζει πάρα πολύ ε, σοβαρό ε, ρόλο και όπως και η κυρία Χάντζικ νομίζω ότι θα συμφωνήσω ότι θα πρέπει να γίνουν μη ελκυστικά τα προϊόντα αυτά για τους νέους. Επίσης ε, η εναρμόνιση ενδεχομένως να δώσει μεγαλύτερη ε, μεγαλύτερο χώρο στα παράνομα προϊόντα. Ε, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο σε χώρες οι οποίες ε, έχουν ήδη εισαγάγει τις εικόνες στην συσκευασία. Υπάρχει και ένα hearing, μια ακρόαση στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος που αναφέρεται ακριβώς ε, στις ε, προστιθέμενες ουσίες αυτές τις πρόσθετες που μπαίνουν στα τσιγάρα και νομίζω ότι και κατά αυτήν την έννοια ε, πρέπει να στηριχτούν ε, οι νέοι έτσι ώστε να αποτραπεί το ξεκίνημα του, του καπνίσματος, να βοηθηθούν οι νέοι και οι λιγότεροι ε, νέοι να σταματήσουν το κάπνισμα. Ξέρω κύριε Πρόεδρε ότι είπατε ότι δεν έχουμε χρόνο, αλλά παρόλα αυτά να πω ότι Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, την ώρα της ε, ακρόασης, έστειλα και κάποια ε, μηνύματα ε, μέσω tweet για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και είχα πάρα πολλές απαντήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν, θέλουν όλοι να καταλάβουν καλύτερα τι είναι αυτό το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δεν υπάρχουν ούτε κανόνες ενίας αγοράς ε, για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πρέπει να το διευθετήσουμε το ζήτημα αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί και η αγορά αυτών των τσιγάρων. Ε, ε, εντάξει, ενδεχομένω αυτά τα τσιγάρα βοηθούν αυτού που θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να κατανοήσουν ότι ακόμα και αυτά τα τσιγάρα δεν είναι καλά για την υγεία. κυρίως ε, δεν να βοηθήσουμε να μην ξεκινήσουν καν με το ηλεκτρονικό αυτό τσιγάρο αυτοί που ε, θέλουν να ξεκινήσουν το κάπνισμα. Θα περιμένω την ε, συνέχεια της συζήτησης και καλωσορίζω αυτήν την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ πάντως από ό,τι κατάλαβα είναι θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει η οδηγία για τα ιατρικά προϊόντα. Κύριο Σμίτ έχει το λόγο. Πρόεδρε, και εγώ θεωρώ ευπρόσθεκτη την οδηγία, όχι όμως σε κάθε τη σημείο. Ουσιώδες πάντως είναι να, δούμε, να βρούμε τρόπους ώστε να αποτρέψουμε την προαγωγή του σιγαρέτου στους νέους. Εγώ κάπνιζα παλιά μου να καπνιστής, είχα ξεκινήσει μάλιστα αρκετά νωρίς και άνθρωποι όπως εγώ συχνά γινόμαστε ακόμη πιο αυστηροί όταν ξεφεύγουμε από το ε, τσιγάρο. Πάντως πιστεύω ότι η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο θα πρέπει με ισορροπημένο τρόπο να χειριστεί το θέμα αυτό. Είναι πολύ ευαίσθητο, διότι εάν σήμερα εμφανιζόταν το κάπνισμα, θα ήταν απαγορευμένο φαντάζομαι θα απαγορευόταν αμέσω. Ίσως λοιπόν κάποιο ο οποίο θέλει να είναι πολύ αυστηρός, ίσω θέλει να φτάσει μέχρι την ολική απαγόρευση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε κάπω πιο μετρημένοι. Αυτό θέλω να πω από πλευρά μου και από τη δική μου σκοπιά, αλλά νομίζω ότι μπορώ να φτάσω μέχρι αρκετά αυστηρές διατάξει προκειμένου να προστατευθούν οι νέοι. Το παράνομο εμπόριο στο, στα τσιγάρα. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τα περισσότερα μάλιστα, η μεγαλύτερη αξία σε λαθρέα προϊόντα είναι αυτή των τσιγάρων με 10 δισεκατομμύρια ευρώ όπως υπολογίζουν οι κυβερνήσεις των κρατών μαρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι χάνουν από το λαθρεμπόριο είτε σε προϊόντα απομίμησης είτε σε λαθρέα τσιγάρα ή προϊόντα καπνού. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο βέβαια με την απώλεια σε έσοδα, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα αυτά, ο τεράστιος όγκο των ελαφρών συναλλαγών, αξιοποιούνται τελικά. Σε τι χρησιμεύουν δηλαδή αυτά τα, τα ποσά. Επίσης, μπορούμε να έχουμε μία λύση ισορροπημένη, δίκαιη και να μην ξεχνάμε ότι και η Ευρώπη δεν είναι η μοναδική περιοχή στον κόσμο. Οι ε, ουσίες οι οποίες δίνουν χαρακτηριστική γεύση δεν πρέπει να επιτρέπονται. Δεν είναι λογικό δηλαδή να έχουμε τσιγάρα με γεύση φράουλας ή πίνια κολάντα ή άλλων κοκτέιλ μερικές φορές πρέπει να σας πω ότι κανείς δυσκολεύεται να είναι φιλελεύθερος ε, σε αυτά τα θέματα. Ο Κέινς ήταν αυτός που έλεγε ότι τελικά όλοι φιλελεύθεροι είμαστε, αλλά ίσως τελικά δεν θέλει να πει κάτι άλλο και να βγει βγήκε έτσι. Τέλο πάντων, κάτι είπε ο κύριο Φόξ από πίσω, δεν ακούστηκε και ο κύριο Σμιτ απαντά. Ναι, ναι, και εγώ αυτό ήθελα να πω, αλλά ίσω να μην είναι τόσο εφιόλογο όσο οι, οι Βρετανοί. Εν πάση περιπτώσει, η εισαγωγή των επιδοτήσεων στα προϊόντα καπνού που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν κάνει από εσά εκεί στην ψηφοφορία που την ψήφισε. Ίσως πρέπει να πείτε ότι δεν, το, δεν τολμάτε να τοποθετηθείτε για την οδηγία αυτή. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε αναφανδόν κατά τις επιδοτήσεις των προϊόντων καπνού. Και τώρα φτάνουμε στο τέλος Ε, βλέπω ένα κενό εδώ στο, ε, στη λογική της Επιτροπής, γιατί το καπνός για ισρόφηση από τη μύτη είναι προϊόν της ιστορικής αγοράς, είτε δεν είναι και άρα ρυθμίζεται από την οδηγία, είτε ανήκει στα κράτη-μέλη αρμοδιότητα. Εν πάση βλέπω κενό. αλλά φαντάζομαι ότι και ο κύριος Έγκστροπ θα αποθετηθεί στο θέμα αυτό. Ε, πάντως την ε, ε, επιτροπολογία, νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να, είμαστε, να αφήσουμε ένα περιθώριο στην επιτροπολογία, αλλά για άλλη μια φορά σας λέω κάτω τα χέρια από τον καπνό για μάσημα, το σνούς, το σουηδικό. Εάν θέλει μια χώρα να κάνει διαφορετικές ρυθμίσεις, δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια ε, παρέκκληση, εθνική παρέκκληση και δεν μπορεί να την αγγίξει κανείς. Ο κύριος Άγκστρομ έχει το λόγο αυτό το ομοιόμορφο πακέτο plain packaging, ε, η απαγόρευση των τσιγάρων, των πολύ λεπτών τσιγάρων slim. Εντάξει, μειώνουμε λοιπόν την ελκυστικότητα της συσκευασία ε, για τους νέους ε, ανθρώπους έτσι ώστε να μην ξεκινήσουν να καπνίσουν εξαιρετικά άψογα. Όμως, όμως, λέει και η Κομισιόν και το λένε και άλλοι, εδώ μιλάμε για την ε, ε, αποτροπή νέων καπνιστών. Τι κάνουμε για αυτούς που καπνίζουν ήδη. Εάν κάποιος είναι θυσμένος στο κάπνισμα, το ξέρει ήδη, το, το γνωρίζει, το καπνίζει. Τι γίνεται με αυτούς. Όσο και αν επιτύχουν αυτά τα μέτρα, θα πάρει 30 χρόνια μέχρι να δούμε μια πραγματική βελτίωση στην ε, δημόσια υγεία του πληθυσμού. Τόσο χρειάζεται για να καθαρίσει ο οργανισμός από το ε, τσιγάρο. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι όλοι έχουμε την υποχρέωση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτού που καπνίζουν να σταματήσουν να καπνίζουν. Γιατί αυτό είναι προπόθεση για οποιαδήποτε βελτίωση ε, της ε, υγείας ε, του κόσμου. Εμείς δεν έχουμε συγκεκριμένες αντιδράσεις σαν πράσινοι. Εγώ λέω τώρα σαν Σουηδός μιλάω, βάζω άλλο καπέλο. Ναι, ίσως μυρίζεστε ήδη προς τα που πηγαίνει αυτό. Ε, δέστε τι γίνεται με το κάπνισμα στη Σουηδία. 28% μέσος όρος καπνίσματος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από 40 μέχρι πολύ χαμηλότερα. Η Σουηδία έχει 13% ε, μέσο όρο καπνίσματος, ενώ ε, ο μέσος όρος είναι 23%, ε, 28% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η επίδοσή μας είναι πολύ καλή. Έχουμε επίσης 50% ε, λιγότερη ε, θνησιμότητα λόγω ε, προβλημάτων και καρκίνου των πνευμόνων από ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να σας δώσω πολλές στατιστικές. Πολλές στατιστικές. Είμαστε στα χαμηλότερα όσον αφορά ε, ε, θανάτους από καρκίνο, πνευμόνων και άλλου ε, είδους. Επομένως η δημόσια υγεία υποφέρει πολύ λιγότερο. Επομένως με αγχώνει λίγο το γεγονός ότι η Κομισιόν αποφάσισε να απαγορεύσει εντελώς τον καπνό για μάσημα, τον σουηδικό σνούς, και πώς να σας το πω. 700.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα από ε, σχετικές με τον καπνό ασθένειες. και αν κατέβαιναν στο επίπεδο της ε, Σουηδίας τότε θα είχαμε 350.000 πρέπει να τα συζητήσουμε, πρέπει να δούμε τα ε, επιστημονικά ευρήματα. Όλοι συμφωνούν βεβαίω ότι το καλύτερο είναι να μην χρησιμοποιήσει κανεί κανένα προϊόν, το καπνού, προϊόν καπνού, κανένα προϊόν που να περιέχει νοικοτήνη. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν κάποιοι να καπνίζουν. Και η, ε, το, το, η σουηδική εμπειρία ε, και η εμπειρία της γυναίκας μου εν προκειμένου κατέδειξε ότι πολλοί κατάφεραν να κόψουν το τσιγάρο χρησιμοποιώντας αυτόν τον καπνό για μάσημα στη Σουηδία, αυτό το σνούς. Και εάν τελικά σταματήσουν να καπνίζουν, αυτό θα είναι πολύ καλό για την υγεία τους και για τη δημόσια υγεία γενικότερα. Συμφωνώ λοιπόν, συμφωνώ με αυτά που λέει η Κομισιόν. Γνωρίζουμε ότι όντως το, το σουηδικό πείραμα ας πούμε έχει πετύχει. Δεν ξέρουμε όταν μεταφερθεί εκτός Σουηδίας εάν ε, θα έχει την ίδια επιτυχία. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο μπορούμε να το αφήσουμε. Ας αποφασίσει η εθνική κυβέρνηση για, αυτές τις, ε, για αυτά τα στοιχεία. Εάν συγκρίνεται τη Σουηδία με την Φιλανδία και την Δανία, εμείς έχουμε ε, το μισό του ποσοστού των καπνιστών, που είναι πολύ κοντινές μας χώρες με πολλά παρόμοια στοιχεία. Και επομένως όλα αυτά συνηγορούν στο να διατηρηθεί ο καπνός για μας στη Σουηδία. Λοιπόν, εάν όλα προχωρήσουν όπως ε, ε, αναμένουμε, τότε λέτε θα μειωθεί το κάπνισμα κατά 2%. Ωραία. Εάν όμως καταφέρναμε να φτάσουμε στο, ευρω... στο σουηδικό επίπεδο θα είχαμε μειώσει το κάπνισμα κατά 15%. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ εύκολο το όλα αυτά. Τώρα, σκιώδες. Υπενθυμίζω όπως ότι τελειώνει ο χρόνος μας. Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να τα συζητήσουμε, αλλά ας ακούσουμε τους σκιώδες και μετά όποιον άλλον αν προλαβαίνουμε. Ο κύριος Μπίλαν έχει το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο σήμερα καλούμεθα να συζητήσουμε και ε, πρόκειται δηλαδή για αυτά τα προϊόντα καπνού. Πρόκειται επίσης για τους κανόνες που θα διέπουν την εμφάνιση των προϊόντων καπνού. Να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για το έργο το οποίο επετέλεσε, γιατί το σημαντικό αυτό θέμα ε, είναι συναρπαστικό, οδηγεί σε συναρπαστική φόρτιση, οδηγεί σε έντονες συζητήσεις και Ξέρουμε όλες αυτές τις ενστάσεις που υπάρχουν ε, έναντι της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να σας επισημάνω εγώ τρία σημεία γιατί όλοι ξέρουμε και όλοι συμφωνούμε ότι το κάπνισμα είναι βλαβερό. Οδηγεί σε πάρα πολύ σημαντικές βλάβες της υγείας αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσον η οδηγία υιοθετεί τους πιο δόκιμους τρόπους για να επιτύχουμε τον σκοπό μας. Να δούμε δηλαδή ποια είναι η πιο σωστή νομοθετική λύση. Εάν τελικά εγκριθεί έτσι όπως είναι η οδηγία θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις για τα κρατη κάποια κράτη-μέλη και θα έχουμε επομένω ε, σε επιπτώσεις και για κάποιους κλάδους ε, της βιομηχανίας και για κάποιες περιοχές, περιφέρειες της Ένωσης. Αυτό να το λάβουμε υπόψη. Τώρα, άλλο θέμα λαθρεμπορία και παράνομη εμπορία. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα ήδη σήμερα. Ε, φυσικά και προσπαθούν, ε, όπως είπαμε, ε, οι... όσοι εμπορεύονται στον αυτά τα παράνομα προϊόντα καπνού να κάνουν ελκυστικό το προϊόν τους. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώ θα δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα σε σχέση με, με, τα απαγορευόμενα προϊόντα, αυτά που θα απαγορευτούν, α πούμε τα, τα τσιγάρα slim. Ε, αν τα απαγορεύσουν αυτά τα τσιγάρα, τότε φοβάμαι ότι θα αναπτυχθεί μια μαύρη, μαύρη αγορά. Ε, ε θα, γίνει, θα γίνει πραγματικός χαμός όσον αφορά τα, την πώληση τέτοιων παρανόμων προϊόντων ε, και μέσω διαδικτύου. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο. Αυτό έχει επιπτώσει στην εσωτερική αγορά, γιατί ο στόχος της οδηγίας TPD είναι να μειώσει τους καπνιστές, ιδίω όσον αφορά τους ε, ανήλικους, τους νέους τέλος πάντων. Αλλά ε, να δούμε μήπως ε, ο σκοπός αυτός δεν επιτυγχάνεται άπαξ και καταστεί εφικτό να διεξάγεται εμπορία προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου. Να δούμε επομένω πώ θα λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε τι λύσει μπορούμε να υιοθετήσουμε και όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη. Και σα ευχαριστώ. Ο Πρόεδρο. Εγώ συνάδελφοι. Θα σα πω ότι έχουμε τρει συναδέλφου οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο. 24 και 25 Απριλίου πάντω θα το ξανασυζητήσουμε. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Εάν έχετε κάτι σημαντικό να πείτε, παρακαλώ κρατήστε το για τότε, για 25 Απριλίου. Αλλιώ, κύριε Μάιερ. Ναι, εδώ μιλούμε για ένα θέμα το οποίο έχει πολλές συνέπειες για τη δημοσιογραφία Είναι ένα θέμα το οποίο όμως ε, ε, στο οποίο πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση των συνεπειών, όπως και το επόμενο που έχουμε στην μέση διάταξη. Λοιπόν, έχουμε δύο φορές εγκρίνει οδηγία για την ε, ε, απαγόρευση διαφήμιση στα προϊόντα καπνού. Η πρώτη φορά ξέρετε ότι απερίφθη από το δικαστήριο γιατί δεν έχουμε αρμοδιότητα για θέματα δημόσιας υγείας. Η δεύτερη χρειάστηκε μια διαφορετική ε, διευκρίνηση του θέματος της διαφήμισης. Δεν αναφέρεται όμως πουθενά η δημόσια υγεία, τα δικαιώματα των καταναλωτών και ερωτώ σε τι θέμα είμαστε αρμόδιοι. Όταν δεν είμαστε αρμόδιοι για την δημόσια υγεία Είμαστε βεβαίω υποχρεωμένοι πάντοτε σε κάθε θέμα, είτε πρόκειται για τον αέρα, είτε πρόκειται για τα αυτοκίνητα, είτε πρόκειται για το νερό, να μεριμνούμε να μην προσβάλλεται η δημόσια υγεία, αλλά δεν μπορούμε να στηρίξουμε ένα νομοθέτημα σε νομική βάση που αφορά τη δημόσια υγεία. Πρώτη αξιολόγηση και δεύτερον, θα συμφωνήσω και με τον Σουηδό συνάδελφο, ότι όντως στα κράτη αυτά στα οποία δεν υπάρχει απαγόρευση είναι μισή είναι μισά τα νούμερα, μισά τα στατιστικά στοιχεία των ε, πραγματικών καπνιστών. Α κοιτάξουμε λοιπόν ψύχρεμα να θεσπίσουμε μια νομοθέτημα πρακτικό και αποτελεσματικό και όχι με συναισθηματικέ ε, φορτίσεις. Ο πρόεδρος, δεν ξέρω αν είναι <laughs> συναισθηματικά τα στοιχεία που έχουμε και η φόρτιση, αλλά ε, χρόνο δεν έχουμε να τα συζητήσουμε τόσο πολύ. Επομένως, είμαστε 12 και 10 και πρέπει να συζητήσουμε την, το, το κείμενο των κυρίων Μάγερ και Γκέμπχαρτ. Συμφωνώ μαζί σας ότι η δουλειά μας αναβαθμίζει την πρόταση Κομισιόν και συμφωνώ ότι εμείς έχουμε αρμοδιότητα την εσωτερική αγορά και η πρόταση, το κείμενο Χάντζλικ, αυτό θα πρέπει να αφορά. Θα το συζητήσουμε οι σκιώδεις ηγητές μαζί σας. Τρεις, τρεις συναδελφούς ζητήσει το λόγο. Στείλτε τις απόψεις σας, πείτε τα. Και όταν συναντήσει η κυρία Χάνζικ με τους σκιώδεις ηγητές, 24 και 25 θα το ξανασυζητήσουν. Τόσα θέματα θα έχουμε για τότε. πρέπει να συζητήσουμε τις τροπολογίες της έκθεσης Γκέμχαρτ Μάιερ. Και τότε να τα ξαναπούμε. Μένουμε εδώ και δίνουμε το λόγο στην κυρία Χάντσλικ. Ελπίζω να έχετε κάποια ένσταση. Πέστε μας για τη διαδικασία κύριε Χάντσλικ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Θέλω να σας ζητήσω κάτι. Είπαμε 24 και 25 Απριλίου θα έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε την πρότασή μου. Γιατί έχω κάποια σημαντικά ζητήματα από την οπτική γωνία της εσωτερικής αγοράς. Και γι' αυτό, Πρόεδρε, θέλω τότε να αφιερώσετε λίγο περισσότερο χρόνο από όσο δώσαμε σήμερα στο κείμενο. Εγώ θα έχω υποβάλει τα κείμενα για μετάφραση και το μεσημέρι της 6ης Μαΐου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. 17-18 Ιουνίου θα γίνει στην ΙΜΚΟ η ψηφοφορία και τον Σεπτέμβριο θα γίνει η συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια. Ελπίζω να έχουμε περισσότερο χρόνο την επόμενη φορά και σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Ιδίω αν θέλετε να συνδυάσουμε πέμπτη απόγευμα. Σήμερα όμως το απόγευμα, μια που λείπουν κάποιοι συνάδελφοι, δεν μπορούμε να έχουμε χρόνο για σας τότε. Οπότε κανονίστε συνάδελφοι να είστε ελεύθεροι πέμπτη το απόγευμα την εβδομάδα των Επιτροπών για να το συζητήσουν. Τώρα κλείνουμε αυτό το σημείο και προχωρούμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων. Έχουμε δύο συνεισηγητές, όπως γνωρίζετε. 300 τόσες τροπολογίες έχουμε που έχουν καταρχήν υποβληθεί και έτσι. Ποιος, ποιος θα μιλήσει. Ο κύριος Μάιερ. Κυρία Γκέμχαρτ θέλετε εσείς να αρχίσετε. Όχι, ο κύριος Μάιερ. Hans-Peter Τελευταία φορά έλαβε το λόγο πρώτη η κυρία θα δώσω το λόγο στον κύριο Hans-Peter Meyer. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Νομίζω ότι η Εύλην και εγώ, όπως θα έχετε διαπιστώσει όλοι, διαφωνούμε απολύτως ως προς την προσέγγιση στο θέμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Ιουνίου του 2011 ολόκληρο το Κοινοβούλιο και κατά πλειοψηφία σαφή υπερψήφισε την ιδέα ενός εκούσιου μέσου. Και το 2013 αποφασίστηκε η οδηγία για την ε, διευθέτηση των διαφορών ODR, ADR. Μέχρι λοιπόν τη θέση εφαρμογή των μέτρων αυτών θα χρειαστεί να περάσει αρκετός χρόνος μέχρι να τον καταλάβει ο εισηγητής, να τον αντιληφθεί. Η ουσία πάντως είναι ότι δεν έχουμε ένα μέσο. Προσπαθούμε με τις ε, εκστατείες ενημέρωσης να δώσουμε την, τα στοιχεία. Χρειάζεται διεύρυνση των δυνατοτήτων, άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς και θα ήθελα να υπογραμμίσω σε τι εξυπηρετεί η παρουσία μας αυτήν εδώ την Επιτροπή. Η αξιολόγηση συνεπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουμε συζητήσει ήδη νομίζω καταλήγει στο ότι χρειάζεται μια νέα προσέγγιση. Και αυτό πρέπει να πράξουμε. Οι επιχειρήσεις συνήθως δεν ε, θεωρούν πρόβλημα ή πρόσκομα στην πώληση στο εξωτερικό την ε, διαφορά γλώσσας. Στα 27 και σε λίγο 28 κράτη-μέλη ε, μπορεί να δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα και να έχουν διαφορούς συνεργάτες που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, αλλά όπως και να έχει νέα γενναία ε, και κυρίως μέσα από το, την επικοινωνία του υπολογιστή και το διαδίκτυο μιλάει πεστρό τα αγγλικά, επομένως πρόβλημα γλωσσικό δεν εμφανίζεται. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι δεν θα είναι το πρόβλημα ως προς την εξυπηρέτηση της ιστορικής αγοράς μακροπρόθεσμα το γλωσσικό. Χρειάζεται πάντως ένα σύστημα ε, για λόγους ασφάλειας δικαίου ασφάλειας για τον επιχειρηματία, για τον πολιτή, για τον αγοραστή, για τον καταναλωτή. Ένα απλό σύστημα το οποίο πιστεύω είναι ικανοποιητικό αυτή τη στιγμή μου φαίνεται ε, το καλύτερο σύστημα αυτή τη στιγμή. Βέβαια ως προς τις ε, ε, επιλογές που μπορεί να προσφέρονται μπορεί να ελεγχθεί το κατά πόσον ισχύει η εκούσια αξιοποίησή τους, το πόσο τα κράτη-μέλη τις σέβονται ή τις προσφέρουν σαν επιλογές. Και κατά πόσον τα όρια που έχουν προσδιοριστεί ισχύουν. Εάν ένα σύστημα εκούσιο επαληθευθεί και μέσα σε 4-5 χρόνια αποδειχθεί ότι λειτουργεί ικανοποιητικά, μπορεί δεν είναι απαραίτητο καταρχά να μείνει σε εκούσια βάση και στο επόμενο διάστημα, αλλά μέσα στην πενταετία μπορεί να επαληθευτεί και να θεωρηθεί ότι είναι ικανοποιητικέ οι διατάξει του και μπορεί να γενικευθεί. Μιλήσουμε μόνο ότι η οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή έχουν φέρει, έχει προσφέρει κάποιες λύσεις και προστασία αλλά όχι όσοι θα θέλαμε, όχι επαρκή. Επί παραδείγματι ορίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής σύναψης μιας σύμβασης, αλλά δεν ε, ορίζει το ουσιαστικό δίκαιο το δίκαιο το σχετικό με τις διαφορές, σε παραδείγματι, το δίκαιο της ε, ανάκλησης της εντολής από 14 ημέρες. Μπορεί να ρυθμίζετε, αλλά δεν ρυθμίζεται το εξάμεινο για την ανατροπή. Επομένως, όταν έχουμε ένα εκούσιο σύστημα μπορούμε πιστεύω να δώσουμε καλύτερες λύσεις για τους καταναλωτές. Οι αθέμητες ε, ρήτρε, ε, τα δικαιώματα στις, στην εγγύηση, τα σχετικά με την εγγύηση, πάλι δεν καλύπτονται και έχουμε να κάνουμε μια ελάχιστη εναρμόνιση, γιατί υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Ε, η αποζημίωση και τα επιτόκια τα σχετικά πάλι δεν ρυθμίζονται. Είναι στο χώρο του εκουσίου, της εκούσιας ρύθμισης. Η προσυμβατική υποχρέωση ενημέρωσης πάλι προβλέπεται μεν, αλλά χωρί καμία κύρωση για το τι συμβαίνει σε περίπτωση παραβίασή τη. Και εδώ χρειάζεται το σχετικό ουσιαστικό δίκαιο ε, να ε, ενταχθεί στην νομοθεσία. Στην ανάκληση πάλι. Υπάρχει αυτή η ευκαιρία, αλλά μπορεί να πει το κράτος μέλος μπορεί να πει ότι υπάρχει δυνατότητα τη ανάκληση στην αρχή τη συμβάσεω, αλλά σε περίπτωση που είναι μία ε, σύμβαση διαφιλονικούμενη, τι συμβαίνει, υπάρχει δυνατότητα τη ανάκληση ή όχι. Όλα αυτά δεν προβλέπονται. Και όταν σε ένα κράτος μέλος προβλέπεται η παραγραφή χρειάζεται όχι η διετία που προβλέπεται στις γενικές διατάξεις, αλλά μια μακρύτερη περίοδος η οποία να προσφέρει επαρκείς εγγύησεις. Όπως είπα, ελάχιστη εναρμόνιση ή μερική εναρμόνιση, πάντως όχι ένας κανονισμός, γιατί ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη θα αντιδράσουν, θα αντισταθούν και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ. Τροπολογίες. Οι τροπολογίες μου είναι και αυτές. Αρκετές θα δείτε. Ζητώ απλουστευμένες δομές, ένα απλό κανονισμό με παράρτημα, μία δομή απλή που να είναι δυνατόν ε, να την ε, διατρέξει κανείς σχετικά γρήγορα, κατανοητή όχι μόνο για τον ειδικό νομομαθή αλλά για τον απλό καταναλωτή. συνέχεια, συνέχιση στις έννοιες, στη χρήση των ενιών και των ορισμών που χρησιμοποιούνται, όχι δηλαδή άλλες έννοιες για το τι σημαίνει καταναλωτής ή επιχείρηση. Μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ των δύο συμβαλωμένων μερών, υψηλό επίπεδο προστασίας φυσικά αλλά και από την πλευρά της επιχείρησης πρέπει να υπάρχει ένα επαρκές περιθώριο λειτουργίας, δράσεως, δεν μπορούμε να περιορίσουμε τελείως, να, δεσμεύσουμε τις επιχειρήσεις. Η ε, παραγραφή, η περίοδος των 10 ετών πρέπει να περιοριστεί στα 6, για να μπορεί και ο πολιτής να κατανοήσει γιατί επιβάλλεται αυτή η διάταξη, να την αποδεχθεί. Και τελειώνω πρώτα σιγά. Εάν κοιτάξετε στο διαδίκτυο, το Amazon ας πούμε ανοίξτε και δείτε πόσες σελίδες βγαίνουν στον ιστότοπο αυτών που δίνουν πληροφορίες για τα συμβατικά δικαιώματα κτλ. Και βέβαια πρέπει να είναι κάτι, ε, γι' αυτό ζητώ να είναι η πληροφορία που θα δίνετε στο διαδίκτυο ευανάγνωστη, σαφής, συνοπτική, κατανοητή. Οι έννοιε, όπω είπα πρέπει να είναι σταθερές, πρέπει δηλαδή η, μία, η κάθε έννοια να αντιστοιχεί σε ένα αντικείμενο, να μην είναι περίπλοκη. Και σε σχέση με το Συμβούλιο θα πρέπει να ε, ε, βρούμε λύσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν δεκτές με το Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή λύσεις οι οποίες ε, απορρίπτονται ανεφετέρου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε κάποιες προτάσεις για τις εξαποστάσεις, ε, πωλήσει, συμβάσεις, ε, με βάση την αρχή της εκούσιας της ε, αποδοχής της, ε, του ε, εκούσιου συστήματος και εφόσον αυτό λειτουργήσει να προχωρήσουμε σε μια γενίκευση όπως είχα πει. Και παραλαμβάνω, η ενιαία αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο σε κάθε μέρος, σε κάθε αγορά. Ε, εάν μπορέσουμε με την οδηγία αυτή να δώσουμε καλές λύσεις για την εσωτερική αγορά, τόσο το καλύτερο. Αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε ποτέ ενιαίες λύσεις για ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Απλώς μπορούμε να προσπαθήσουμε να ε, παραμερίσουμε εμπόδια τα οποία παρεμποδίζουν την ε, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος και η συνεισηγήτρια κυρία ε, Γκέπχατ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα εγώ έχω μόνο 10 λεπτά, τι να κάνω. Ε, ένα τεταρτάκι και μίλησες. Εν πάση περιπτώσει. Με το Hans Πέντερ συμφωνώ σε ένα θέμα ότι διαφωνούμε. Είναι το μόνο σημείο σύγκληση μεταξύ μα. Όντω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πει σε ένα ψήφισμα του ότι θα πρέπει το εκούσιο σύστημα να εξεταστεί ω λύση, αλλά ταυτόχρονα με μία αξιολόγηση συνεπειών που ήταν συνδεδεμένη μαζί του και η οποία θα δίνει ε, πιστικά επιχειρήματα ότι είναι όντως το καλύτερο μέτρο αυτό. Και έτσι ε, ότι καλύπτονται οι ανησυχίες και των επιχειρηματιών και των καταναλωτών. Και πρέπει να σας πω, ξεκινώντας, ότι δεν ε, το ε, αντιμετώπισα το θέμα αυτό ελαφρά την καρδία. Έκανα αμέτρητες συνομιλίες με καταναλωτές και οργανώσεις καταναλωτών, αμέτρητες επαφές με επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οργανώσεις επιχειρηματιών και η μεγάλη, μεγάλη, πολύ μεγάλη πλειοψηφία μου είπε μας δυσκολεύει αυτή η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής το καθεστώς αυτό, το εκούσιο με 28 κράτη, μας δυσκολεύει πολύ, με 28 μέλη καλύτερα. Και γι' αυτό ζητώ να επαρελθευτεί η αξιολόγηση επιπτώσεων με τα συμπεράσματα που έχουμε Δεν έχω πολύ χρόνο, όπως είπαμε, θα το διατρέξω κάπως γρήγορα, διαβάστε και στις πιο αναλυτικά. Τώρα, γιατί έχουμε αυτό καθεστώς με 28 μέλη, να σας πω. Γιατί ε, το σύστημα αυτό θεωρητικά δεν είναι εφαρμόσιμο με 27-28 κράτη-μέλη. Η μείωση ε, του κόστους είναι μη το βλέπετε και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σελίδα 117 ε, της μελέτης αξιολόγησης. Δεν είναι αυθαίρετα δηλαδή τα στοιχεία που σας προσφέρω. Και ξέρετε, με απασχόλησε πολύ το τι θα κάνω από τη στιγμή που διαπίστωσα ότι δεν ε, λειτουργεί το σύστημα αυτό και αφού τόσοι πολλοί ε, επαγγελματίε ε, και ενδιαφερόμενοι του χώρου μου είπαν δεν το θέλουμε συμφωνούμε με τον Χάνς Πέτερ ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος χειρισμού της υπόθεσης. Δηλαδή υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία μπορούν να εξοικονομηθούν ούτως υπήσιν από την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Και ακριβώς τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν εδώ είναι... Ο ε, ότι η επιλογή της πλήρους εναρμόνισης λόγω της αντίδρασης του Συμβουλίου απέτυχε, αλλά θα πρέπει να πούμε, να μην ξεχάσουμε να πούμε, ότι μια ανασχετική μειονότητα ήταν αυτή του Συμβούλου, η οποία τάχθηκε κατά του εκούσιου συστήματος, ε, ότι υπάρχει μια ε, ανασχετική μειονότητα και κατά του συστήματος του εκούσιου στο σύστημα, άρα ίσως ούτε αυτό να μην λειτουργήσει. Και άρα θα πρέπει να διαρωτηθούμε ποιον δρόμο θα επιλέξουμε. Αν δεν έχουμε ούτε την πλήρη εναρμόνιση, ούτε το κατεπιλογήν σύστημα, και με την οδηγία των, για τους καταναλωτές ε, έχουμε επιλέξει, ξέρετε με τον Ανδρέα Σφάπ, την, ε, το δρόμο της ελάχιστης ή κάθετος και μικτής εναρμόνισης. Μήπως αυτό είναι η καλύτερη ευκαιρία που θα είχαμε να περάσει ένα σχετικό νομοθέτημα, γιατί εκεί και ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας μπορούν να ενστερνιστούν το εγχείρημα και να μας βοηθήσουν και σε σχέση με κάποια εμπόδια προς κόμματα, αντιδράσεις και αντιστάσεις που μπορεί να έχουμε σε επίπεδο Συμβουλίου. Άρα ίσως θα πρέπει να αναστήσουμε έναν ελεκτικό δρόμο. Στην οδηγία δηλαδή για την προστασία των καταναλωτών, αυτό που ε, ήταν ο λόγος της αποτυχίας των προσπαθειών μας ε, σε επίπεδο συμβουλήτων ότι δεν ήθελαν ε, εναλλακτικέ. Τώρα, ε, εναλλακτικέ τι σημαίνει, ότι δεν λειτουργεί το σύστημα σε πλήρη εναρμόνιση, δεν λειτουργεί το σύστημα το εκούσιο, δεν γίνεται αποδεκτό δηλαδή. Άρα κάποια εναλλακτική πρέπει να προτείνουμε και στρέφομαι και πάλι, μάλλον θα αναφέρω και πάλι τον κύριο Σφαπ. Τι κάναμε, Αντέγραψα ούτως ή από τον κύριο Σφάπ, από τη δουλειά αυτή που είχαμε κάνει και καταγράφω σε έναν πίνακα το πώς ε, βλέπω αυτές τις εναλλακτικέ. Στην ε, Οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή, ευχαριστώ Ανδρέας, είχαμε βγάλει τον τίτλο αυτόν περί οριζόντιας οδηγίας και προχωρήσαμε κατακόρυφα και μιλούσαμε για ελάχιστες ε, νόμιμες ε, εγγυήσεις για την παροχή υπηρεσιών κτλ. Έτσι λοιπόν και στις τροπολογίες τις οποίες εγώ επεξεργάστηκα ακολούθησα την ίδια μέθοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, συμπεριλάβει στην πρότασή της πολλές θέσεις τις οποίες εγώ βρίσκω θετικές και προσπαθώ να συμπεριλάβω. Δεν μου φαίνονται όλες οι προτάσεις της Επιτροπής δηλαδή εσφαλμένες, απλώς η προσέγγιση είναι το πρόβλημα στην υπόθεση αυτή, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε δηλαδή, και προσπαθώ μέσα στο νέο μου σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σουάπ. Εύελιν, με συγχωρείς. Χρειάζομαι και χρόνο για τους σκιώδεις, έτσι, αυτό πρέπει να σου πω. Και μας έχουν δώσει 10 λεπτά ακόμα οι διερμηνείς, αλλά... Ναι, εντάξει, μάλλον χρειάζομαι περισσότερο χρόνο για να παρουσιάσω την ε, θέση μου. Δεν ήθελα να σε κόψω, αλλά παρόλα αυτά ο χρόνος λείπει. θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο βέβαια, αλλά να έχουμε μία πρώτη ανταλλαγή και ευχαριστώ του διεμηνείς που μου δίνουν λίγο χρόνο. Shadow Medium, Public Procurement. I will follow later on, Mr. Also, wir sind uns hier einig, wir haben, wir haben zwei Entwürfe. Ναι, εντέλει ο κύριος Κρότσμαν, ελάτε. Λοιπόν, έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, δύο διαφορετικές προτάσεις για το ίδιο θέμα και πρέπει να ε, δούμε πώς θα το χειριστούμε. Εδώ έχουμε διαφορετικές νομικές παραδόσεις και νοοτροπίες στην Ευρώπη ως προς τα δικαιώματα του καταναλωτή και πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί, ποιο πρόβλημα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Ε, το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί επαρκώς το διαδικτυακό ή το εξαποστάσεως εμπόριο μέσα στην εσωτερική αγορά. Ε, διότι θέλουν και τα μικρότερα και οι καταναλωτές από μικρότερα κράτη ή μικρότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για ε, να παραγγείλουν εξ αποστάσεως ένα προϊόν, εφόσον όμως γνωρίζει και τι είδους ε, δικαιώματα έχει ο καταναλωτής. Αν θέλει ένας Μαλτέζος να παραγγείλει ένα προϊόν από την Γερμανία, πρέπει να γνωρίζει τι συνέπειες έχει αυτή η προσέγγιση του και αυτή η πράξη. Ο κύριος Μάιερ. προσπαθεί να δώσει λύσεις οι οποίες να προσφέρουν βέβαια καλύτερες λύσεις για τον καταναλωτή. με ισορροπημένη όμως προσέγγιση μεταξύ συμφερόντων του πολιτή και συμφερόντων του καταναλωτή. Για να θέλουν και οι πολιτές να εμπλακούν στην ε, περιπέτεια αυτή. Το καθεστώς λοιπόν αυτό των 28 εμπλεκομένων θα υπάρχει εφόσον ο πολιτής και ο καταναλωτής αναπτύσσουν αυτές τις εμπορικές δραστηριότητες και εάν μπορεί ένας πολιτής της Γερμανίας να πολύ με βάση το γερμανικό δίκαιο ε, στη Γαλλία, τη Μάλτα αλλά και στη Γερμανία και να μπορεί να γνωρίζει και αυτός αλλά και ο αγοραστής τι ισχύει. Ο κύριος Μάγερ είπε πολύ σωστά ότι πρέπει να ε, απλουστευθεί η ε, ορολογία Οπωσδήποτε χρειάζεται να πισχναστεί όλη αυτή η ενιολογία και η ορολογία που υπάρχει προς το καλό του καταναλωτή για να είναι πιο ευανάγνωστες διατάξεις. Ξέρουμε, το είπατε και εσείς κυρία Γκέμπχαρτ, ότι δεν θα συμφωνήσετε στην προσέγγιση σας, έχετε τελείως διαφορετική προσέγγιση, αλλά από την άλλη μην ξεχνάμε ότι έχουμε έναν στόχο Και έχει πει ο κύριος Χάνς Πέτερ Μάιερ και ο κύριος Σφάπο ότι είναι πολύ διαφορετικά τα ε, δίκαια, οι ε, παραδόσεις ε, του δικαίου στα κράτη-μέλη. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε μόνο το επιρωτικό δίκαιο, έχουμε και το δίκαιο το σαξονικό. Είναι πολύ διαφορετικέ λοιπόν οι διατάξει και δεν είναι δυνατόν να επιδιώξουμε την αναρμόνισή του. Αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε μια ευκαιρία και να εξασφαλίσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στην αγορά για τον καταναλωτή, για να μπορεί να, να ε, ε, εμπλέκεται σε τέτοιου είδου συναλλαγέ. Μια εμπειρία λοιπόν θα έλεγα πάνω απ' όλα που θα πρέπει να διευκολύνουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριο Φόξ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, η πολιτική μας ε, η ομάδα και εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η νέα αγορά για τον κόσμο, για τις ε, επιχειρήσεις, όμως δεν ξέρω αν είναι προς αυτό το, το, το δίκαιο των πωλήσεων όπως βλέπετε και έχουμε και αυτή το, το health check, τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας αυτής της μελέτης επιπτώσεων και με επιφυλακτικό και όσον αφορά ε, την έκθεση της Επιτροπής. Ήδη είπαμε ότι έχει πολλά κενά, το συζητήσαμε και είπαμε ότι οι εξοικονομήσεις ε, είναι λάθος. Επηρεάζεται των συμβαλωμένων η συμπεριφορά, είπαμε, και επομένως, κατά τη γνώμη μου, αυτή η μελέτη επιπτώσεων ε, είναι μεροληπτική. Δηλαδή, είναι φτιαγμένες, κομμένοι και ραμμένοι για να ε, πετύχει το στόχο της η Επιτροπή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Κρότσμαν, ο κύριος ε, Μέιερ ε, είναι σεβαστοί, όμως από ό,τι είπανε, δεν έχουμε ένα κοινό νόμο τόσο ώστε να άρουμε τους φραγμούς του εμπόριου. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν αυτό το οποίο είπατε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε τρία διαφορετικά νομικά συστήματα, ένα για Αγγλία και Ουαλία, ένα άλλο για Σκοτία και ένα άλλο για την Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό δεν εμποδίζει το εμπόριο μεταξύ αυτών των τριών περιοχών καθόλου. Και κατά την άποψή μου, το να πείτε ότι αποτελεί φραγμό στο εμπόριο ε, τα διαφορετικά συστήματα ε, είναι μια πρόφαση για να πετύχετε περισσότερη και τον ρύθμιση στην Ευρώπη, το οποίο είναι θεμητό στόχο, αλλά είναι ανακριβέ να λέτε ότι υπάρχει τέτοιο φραγμό στο εμπόριο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η κυρία Γκέφχαρτ είναι πιο πρακτική, η προσέγγισή της είναι πιο λογική και επομένως όσον αφορά την αλλαγή, την τροποποίηση της, ε, της, της, της, της, της ε, ε, πρώτης κομισιόν θα, θα την ε, ψηφίσουμε. Θα έχω κι άλλα να σας πω, νομίζω ότι θέλετε να τα ακούσετε. Κυρίε και κύριοι, λέει ο Πρόεδρος. Λυπάμαι. Βάλαμε πάρα πολλά θέματα. σήμερα το πρωί. Πάντοτε, πάντοτε πέμπτη πρωί υπάρχει πίεση είχαμε και τις ψηφοφορίες. Οπότε αν μπορούσατε να έρχεστε πέμπτη απόγευμα θα τα πηγαίναμε μεγαλύτερα Τέλος πάντων. Αξιόλογη συζήτηση. Και συνούμε με τη γραμματεία για το πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε, να διαχειριστούμε τις τροπολογίες γιατί όλοι, όπως ο κ. Φόξ, θέλει να τροποποιήσει την πρόταση Γκέμπχαρτ Πάρα πολύ χρήσιμα τα όσα προτείνει η κυρία Γκέμπχαρτ. Θα τα βρουν οι συγητές με τους σκιώδες συγητές. Δεν έχουμε χρόνο. Και δεν θα δώσει άλλον το λόγο, θα τα πούμε την επόμενη φορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. προθεσμοί για τροπολογίε 23 Απριλίου και θα συζητούν τροπολογίες 29 και 30 Μαΐου. Και θα πρέπει να δούμε γιατί θα γίνει και θα συζητηθούν οι συμβαστικέ τροπολογίες και αυτό ίσω είναι, ίσως αυτό αλλάξει τα πράγματα. Θα ψηφίσουμε στι 9 Ιουλίου, τέλος πάντων θα το ξανασυζητήσουμε. Οπότε ίσως αλλάξει το χρονοδιάγραμμα. Να δούμε τι θα πει η νομική επιτροπή. Αλλά βέβαια θα πρέπει να συζητηθεί όντω και η πρόταση Γκέμπαρτ. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω, έχετε να πείτε κάτι τελευταίο, κυρία Γκέμπαρτ και κύριε Μάγερ. Όχι. Όχι, κυρία Γκέμπαρτ. Ναι, Πρόεδρε. Απλώς θα παρακαλέσω να μην μας βάλετε στο, στη σειρά μετά τον το καπνό την επόμενη φορά στην ημερήσια διάταξη. Ναι, ναι, λέει ο Πρόεδρο, αλλά ξέρετε, χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο για το απόγευμα. Μία ώρα θα μα περισσέψει το απόγευμα, γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε ηγητέ που θα έρθουν. Κύριε Πέτερ Μάιερ, όχι. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ του Ερμηνεί, λέει ο Πρόεδρο, που μα έδωσαν χρόνο. Θα τα πούμε στι τρει. με τρεις ακόμη εκθέσεις πολύ ενδιαφέρουσες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά με τον κύριο Χάνς Πέτερ Μάιερ και πάλι και άλλα θέματα. Θα προγραμματίσουμε λοιπόν όσο πιο καλά μπορούμε και τις προσεχείς επαφές. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλά μας στις